Colleagues, start. not here, Λοιπόν, συνάδελφοι, θα ξεκινήσω γιατί έχουμε και δύο ψηφοφορίες και μία ακρόαση και δεν θέλω να καθυστερήσουμε γιατί έχει ζητήσει και η κυρία Κούνεβα, η Επίτροπος, να έρθει και να μιλήσει στην αρχή της ακρόασης. Έχετε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Δεν έχω κάποιες ιδιαίτερες ανακοινώσεις. Ήθελα απλά να, ρωτη... να ζητήσω από τον κύριο Μλάντενοφ να μας πει λίγα λόγια για την ε, αποστολή στην Βουλγαρία για να ενημερώσετε τους απόντες. Βεβαίω, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους που ήρθαν τελικά στην αντιπροσωπεία και τη γραμματεία για την οργάνωση. Είχαμε, κάνουμε αρκετές ενδιαφέρουσες ε, επισκέψεις. Ε, πρώτα απ' όλα συναντηθήκαμε με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Οικονομικών Υποθέσεων του Βουλγαρικού Κοινοβουλίου. Πήγαμε στο Υπουργείο Οικονομικών, είχαμε συναντήσεις ε, με οργανώσεις καταναλωτών και επιχειρηματιών. Πήγαμε στο Πλοβδίβ, μια πόλη ε, ανατολικά της ε, Σόφιας ε, και συναντηθήκαμε και με αρκετά επιμελητήρια. Δύο βασικά ήταν τα θέματα. Πρώτα απ' όλα η ενεργειακή ασφάλεια. Όπως ξέρετε η Βουλγαρία ήταν η χώρα η οποία υπέφερε περισσότερο κατά την κρίση με το φυσικό αέριο με τη Ρωσία. Οπότε πολύ συζητήσαμε για αυτό το θέμα, πρόσβαση στο αέριο, καθώς και πυρηνική ενέργεια και δεύτερον η οδηγία των υπηρεσιών και η μεταφορά του βουλγαρικού δικαίου. Οι οργανώσεις των καταναλωτών έδειξαν κάποια ζητήματα, πρώτα απ' όλα το ότι λαμβάνουν περιορισμένη χρηματοδότηση ακόμα για τις δραστηριότητες τους. Βεβαίως αυτό συζητήθηκε γιατί κάποιοι λένε ότι χρειάζονται περισσότερη χρηματοδότηση, άλλοι θα έλεγαν πως οι οργανώσεις των καταναλωτών θα έπρεπε να μπορέσουν να είναι αυτόνομες, να μπορούν να είναι αυτόνομες. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγους μήνες ε, είχαμε ακούσει αυτές τις οργανώσεις των καταναλωτών από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και είχε ακουστεί τότε μια ιδέα για να δούμε πώς μπορούν να συνεργαστούν αυτές οι οργανώσεις για να μοιραστούν τη γνώση τους κτλ. Ίσως στην επόμενη θητεία θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να το δει αυτό στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Οι επιχειρήσεις μίλησαν εκ μακρόν για διάφορα ζητήματα διοδότησης, ε, ρυθμιστικά ζητήματα που εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα στις δραστηριότητές τους και κάποια από αυτά τα ζητήματα μάλιστα καλύπτονταν από την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, η οποία είναι κυρίως αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων Υπουργείων βεβαίως. Ήταν λοιπόν μια καλή επίσκεψη θα έλεγα. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουν μαζί μου οι συνάδελφοι πως ε, πραγματι είδαν πως υπάρχουν αρκετές προκλήσεις. Συναντηθήκαμε και με την τοπική αυτοδιοίκηση να δούμε πώς λειτουργεί ιδιαίτερα στην προστασία των καταναλωτών και να δούμε και τις... Ε, να δούμε πώς λειτουργεί το τοπική και στη Σόφια και στο Πλόβντιβ. Πράγματι κάποια ζητήματα όντως μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εξέταση ίσως και μιας νέας ε, επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν ε, να ασχοληθούμε με το επόμενο θέμα, ανάκληση οδηγιών περί μετρολογίας. Θα ήθελα να ρωτήσω το Συμβούλιο. Υπάρχει κάποιος εδώ παρόν. Ο κύριος Βότοπαλ. Ναι, έχετε τον λόγο. I'm glad. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, θα σας δώσω πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου που είχε δύο συζητήσεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και η συζήτηση ήταν κάπως συγκεκριμένη διότι τα διάφορα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές προτιμήσεις για διαφορετικές οδηγίες οι οποίες πρέπει να καταργηθούν και γι' αυτό ζήτησε, ε, ζητήθηκε η γνώμη των επιτετραμένων για καλύτερη νομοθεσία και για νέα ρύθμιση και ελπίζω ότι θα υπάρξει μία νέα πρόταση. Η συνεδρίαση αυτή ήταν την Παρασκευή και τα βασικά χαρακτηριστικά είναι να καθυστερήσει η ημερομηνία εφαρμογής μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2014 που είναι μακρινή ημερομηνία αλλά θα μπορέσει να μας επιτρέψει ε, να καταρτήσουμε νέα οδηγία για τα όργανα μέτρησης και ιδίως για τα παραρτήματα της οδηγίας που χρειάζονται ακόμη. Ουσιαστικά η συζήτηση δεν έδειξε να χρειάζεται οποιαδήποτε από αυτές τις οδηγίες και τα κράτη-μέλη ε, δεν αφισβητούν τα αποτελέσματα της ε, αξιολογήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως σας είπα η συζήτηση ήταν κάπως συγκεχημένη αλλά ήρθαν οι επιτετραμένοι στην τελευταία συνέδριαση και είπαμε ότι θα πρέπει να καταργηθούν αυτές οι οδηγίες και να υπάρξει καλύτερη Κατόπιν αυτού το Συμβούλιο θα διατυπώσει μία τελική θέση εντός των επομένων δύο-τριών εβδομάδων. Ευχαριστώ. Όπως είπατε είναι αρκετά συγκεκριμένο γιατί είπατε ότι από τη μία πλευρά τα κράτη-μέλη δεν χρειάζεται να δουν πώς θα λειτουργήσει ε, η, οδηγία και από την άλλη πλευρά όμως συγχρόνως θέλουν να καθυστερήσουν την πρόταση. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να το διευκρινίσει. Νομίζω πάντως ότι θα πρέπει να το δουν οι συντονιστές και να μας πούν πώς θέλουν να προχωρήσουν. Ο κύριος θέλω να επιβεβαιώσω αυτό που σας είπε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου διότι όντως στην περασμένη Παρασκευή την τελευταία στιγμή έπεσε μια ιδέα από πλευρά της Τσεχικής Προεδρίας να υπάρξει μια συμβιβαστική λύση μέσω μιας δηλώσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα πει ότι δέχεται να καθυστερήσει εφαρμογή και να αξιολογήσουμε πότε θα χρειαστεί να αξιολογήσουμε μέχρι τον Απρίλιο οπότε η Επιτροπή πρέπει να καταρτήσει μία έκθεση να θίξει και το θέμα αυτό, δηλαδή αν υπάρχουν προβλήματα στην αργοεράπη. Κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται όμως, αλλά οτιδήποτε υπάρξει θα συμπεριληφθεί και αυτομάτως θα υπάρξει επίσημη κατάργηση αν ακόμη το σύστημα αυτό ισχύει μέχρι το 2014. Άρα όλα αυτά γίνονται με την επιφύλαξη ότι υπάρχει εσωτερική συνεννόηση και στην Επιτροπή Εσωτερικών Σχέσεων την Παρασκευή θα μπορέσουμε να καταλήξουμε ε, σε μία συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το Κοινοβούλιο πριν ε, διαλυθεί αν συμφωνείτε και να ακολουθήσουμε τη διαδικασία που πρότεινε αυτή η ε, πρόταση και να ακολουθήσουμε αυτή την πρόταση μεταφέροντας την ημερομηνία. Σας ευχαριστώ. Κυρία Γκέπχαρτ, θέλετε κάτι να πείτε? θα πρέπει ούτως ή άλλως να πάει στους συντονιστές. Δεν θέλω να γίνει μια μακριά συζήτηση από αυτού. Έχω όμως μια ερώτηση, διότι υπάρχουν διάφορα πράγματα που έφτασαν στα αυτιά μου σχετικά με ε, τις, τους κανονισμούς και τις οδηγίες που σημαίνουν πλήτη εναρμόνιση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό σημαίνει ότι εάν καταργηθούν αυτοί οι κανονισμοί ε, θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές μετρήσεις στα κράτη-μέλη και θα υπήρχε μία ασφάλεια. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας απαντήσει από αυτού. Δηλαδή ποια θα είναι η επίπτωση αν υπάρξει μία κατάργηση αυτών των οκτώ οδηγιών και ιδίως ε, εάν σταματήσει θα σταματήσει η πλήρης εναρμόνιση την οποία έχουμε επιτύχει σε αυτό το τομέα. Θέλετε να απαντήσετε πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα πιστεύουμε και συμπεριλαμβάνεται στην πρότασή μας ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα εμπόδια διότι ε, ε, οι, τα οχτώ θέματα που καλύπτονται από τις οδηγίες καλύπτονται από διεθνείς προδιαγραφές και έτσι θα συνεχίσουν να ισχύσουν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει κανένα πρόβλημα διότι όπως ξέρετε τα περισσότερα κράτη μελη δεν χρησιμοποιούν καν τις συγκεκριμένες οδηγίες. Δηλαδή είναι οδηγίες που χρησιμοποιούνται ελάχιστα και γι' αυτό πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Αλλά για να υπάρχει μία δικλίδα ασφαλείας θα θέλαμε ε, βάσει των εκθέσεων που θα υποβληθούν από τα κράτη-μέλη μέχρι του χρόνου αν ακόμη υφίστανται προβλήματα οπότε στην έκθεσή μας το 2011 να μπορούμε να επανέλθουμε με προτάσεις. Αλλά δεν νομίζω θα συμβεί κάτι τέτοιο. Όλα αυτά καλύπτονται από διεθνείς προδιαγραφές και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν προβλήματα μέχρι τούδε. Δεν θέλω να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι είναι ασαφές το τι γίνεται με αυτήν την ανάκληση οπότε δεν θέλω να γίνει ε, διαδικαστικό θέμα. Ευχαριστώ τον κύριο Ορτούν για το Συμβούλιο που μας ενημέρωσε και θέλω πρωτού πάμε στις ε, τις ε, ψηφοφορίες να μας παρουσιάσει την έκθεσή του ο κύριος Χάρβορντ για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι το αποτέλεσμα της, του τριμερούς ε, ε, διαλόγου με το Συμβούλιο και των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. θα ήθελα για να σας υπενθυμίσω κάποια πράγματα να πω τα εξής. Όντως, η κοινή θέση της Συμβουλίου δεν μας έγινε γνωστή στις 19 Φεβρουαρίου. Για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν τη διαδικασία δεύτερης ανάγρασης ήταν για μένα απαραίτητο να έχω το έγγραφο αυτό για να μπορέσω να συμπεριλάβω κάποια θέση στην έκθεσή μου και αυτό ακριβώς έκανα. Τώρα, από τότε που πήραμε τα σχόλια της κοινή θέση, πρέπει να πω ότι είχαμε διάφορες συναντήσεις με την Προεδρία του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένη και μία ε, συνεδρίαση με την ε, Γαλλική Προεδρία, προηγουμένως και τώρα με την Τσεχική. Πρέπει να πω ότι όλο το πακέτο είναι πολύπλοκο και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα υπάρξει κανένα κομμάτι το οποίο θα χωριστεί. Όλη η διαδικασία θα ακολουθηθεί ε, από κοινού με τις άλλες εκθέσεις και παραλλήλου με αυτές τους Μέχρι σήμερα, στο κέντρο των διαπραγματεύσεων του Συμβουλίου, το μέλημα ήταν να έχουμε καλύτερη ε, καλύτερη νομοθεσία στα πλαίσια αυτών των οδηγιών. Εμείς πρέπει να πω ότι με την τσεχική Προεδρία δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε, γιατί δεν παρουσιάστηκαν στις δικές μας τροπολογίες συμβιβαστικέ. Πιστεύω ότι και μπορεί να γίνει μετά το γνωστή της εκθεσής μας. Τώρα, στο περιεχόμενο της εκθεσής μας, σε μεγάλο βαθμό, υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν από την Επιτροπή μας μετά τις συζητήσεις πέρσι και δεν υπάρχουν στην κοινή θέση. Υπάρχουν κάποιοι τομείς, λίγοι τομείς, του οποίους με την ε, συμφωνία των ε, σκιωδών εισηγητών έχω κάνει αναδιατυπώσεις και θα ήθελα κυρίως να πιστήσω την προσοχή σας στο θέμα της προστασίας της δυτικής ζωής αυτής της οδηγίας. Αν θα πω ότι είχαμε πρώτα όλα ε, δύο διαφορετικέ δουλειέ. Προστασία τη ιδιωτική ζωή και μετά τα δίκτυα υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στην προστασία ιδιωτική ζωή πρέπει να πούμε ότι προχωρούμε περισσότερο από ό,τι θέση του ιδίου, κυρίω όσον αφορά τα θέματα των κοινοποιήσεων σε περίπτωση που καταστρατηγεί αυτό το δικαίωμα των καταναλωτών. Εκεί που έχουμε προχωρήσει και θέλω να σας πω ότι έχω συνεργαστεί πάρα πολύ με τον κύριο Άλβαρο, με τους δικούς του ε, σκιώδεις εισηγητές για να έχουμε κοινή θέση. Παρόλο το γεγονό λοιπόν ότι προχωρήσαμε πολύ, νομίζω ότι θα πρέπει, επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, να έχω τη συμφωνία όλων δεδομένου ότι πρόκειται, επαναλαμβάνω, για ένα θέμα. Ε, πάρα πολύ ευαίσθητο. Ο κύριος Άλβαρο και οι δικοί του σκιώδεις ηγητές ήρθαν μαζί μου όταν είχαμε τον διάλογο μεταξύ τριών. Έχουμε ένα σετ προτάσεων για το θέμα αυτό των βιβλίο θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή διότι μας βοήθησε όσον αφορά αυτό το αναθεωρημένο κείμενο για να μπορέσουμε τελικά να καταλήξουμε συμφωνία. Πρέπει να πω ότι το πεδίο εφαρμογής της πρότασής μας είναι επίσης ε, κάτι σημαντικό. Θα πρέπει εδώ να συμπεριλαμβάνονται στοιχεία τα οποία μεταφέρονται μέσω των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Όπω πράγματα που αφορούν επισωτικέ κάρτη οτιδήποτε. ή πιστοτικές κάρτες ή οτιδήποτε. Πία, αυτή τη στιγμή δεν ε, περιλαμβάνονται. Αυτό πιστεύουμε ότι δεν είναι σωστό, γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να υπάρξει πρόοδος, ώστε όπως είπα να περάσουμε όλα αυτά όλα μαζί. Ένα άλλο σημείο το οποίο θέλω πίσω την προσοχή σας είναι ένα εντελώς νέο στοιχείο και αφορά τον ορισμό της ε, καθολικής υπηρεσίας. Κάποιες χώρες προσπαθούν να επεκτείνουν όλες τις διατάξεις για να μπορέσουν να συμπεριλάμβουν και τις τεχνολογίες τευριζωνικές. Η Επιτροπή πρέπει να πω ότι έχει καθυστερήσει στο θέμα αυτό των διαβουλεύσεων για το θέμα αυτό. Και αυτό είναι απογοητευτικό. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα μπορέσουν να ληφθούν υπόψη τα πορίσματα των διαβουλεύσεων του στην οδηγία αυτό. Ελπίζουμε ότι θα γίνει περαιτέρω λοιπόν αναθεώρηση το 2010 ε, των ε, οδηγίες ειδικά με, ε, με την καθολική υπηρεσία και Νομίζω ότι για να μπορέσουν να υιοθετηθούν νέες πολιτικές θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Σε μία νέα ε, παράγραφο θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε και κάποια νέα στοιχεία του ορισμού όσον αφορά τις ευρωκοινωνικές ζώνες. Εάν συμφωνήσει το Συμβούλιο, είναι νέο σημείο πρέπει να πω ότι δεν συμπεριλαμβάνονταν στην δεύτερη ανάγνωση, εάν το επιτρέψει το Συμβούλιο μέσω των ε, τροπολογιών πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το προσθέσουμε αυτό σαν νέο στοιχείο και πρέπει να πω ότι υποτελεί την τροπολογία της ε, έκθεσης. Λοιπόν, αύριο θα συναντήσω όλους τους και εισηγητές για να τους ενημερώσω, να δούμε ποια θα είναι η διαπραγματική μας προσέγγιση και τακτική. Ε, σχεδιάζεται νέος διάλογος μεταξύ των τριών στις 4 Μαρτίου και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις φαντάζομαι ότι δεν θα μπορέσουμε να έχουμε όλο το χρόνο που χρειαζόμαστε για τη διαπραγμάτευση. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να σας πω ότι ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν και ξέρουμε ότι θα γίνει σωστά η ψηφοφορία στην Επιτροπή και θα συνεχίσουμε περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις ώστε να μπορέσουμε να γνωμοδοτήσουμε έτσι όπως μας έχει ζητηθεί στα πλαίσια αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Χάρπορ. Ήταν πάρα πολύ εμπεριστατωμένη η εξήγησή σας. Καλό είναι που μας ενημερώνετε για την πρόοδο που επιτυγχάνετε. Πιστεύετε ότι πρέπει να καλέσουμε τον κύριο Ρότφορ, θεία της Επιτροπής. Ας δώσω το λόγο λοιπόν στην Επιτροπή. Σύντομα, παρακαλώ. Δεν θέλω να ανοίξουμε συζήτηση, δεδομένου ότι πρέπει να αρχίσουμε την ψηφοφορία στις 3.30. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν καλωσορίζει το έργο του κυρίου Χάρμπορ στην πρώτη ανάγνωση και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια. Όπως και το, ότι το, γεγονό, το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να θέλει συμφωνία στη δεύτερη ανάγνωση και θα καταβάλουμε και εμείς κάθε προσπάθεια για να το υποστηρίξουμε. Καλωσορίζουμε επίσης ε, πολλά από τα στοιχεία της έκθεσης του κυρίου Χάρμπορ που έχετε μπροστά σας. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Απλά να απαντήσω πολύ γρήγορα στα δύο σημεία που ανέφερε ο κύριος Χάρμπορ για το πεδίο εφαρμογή της ε, ειδοποίησης παράβασης δεδομένων. Εκεί πέρα η κυρία Ρέντινγκ είπε πως αντιλαμβάνεται πλήρως τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου και δεσμεύεται να εξετάσει τρόπους ε, ώστε να διασφαλίσει ότι το σχετικό μέσο θα τροποιηθεί καταλήλως. Για το δεύτερο σημείο, δηλαδή το εύρος της ε, καθολικής ε, παροχής υπηρεσία. Εμείς ε, από την αρχή της συζήτησης θεωρούσαμε πως έπρεπε να συζητήσουμε πλήρως ε, το θέμα αυτό και οποιαδήποτε αλλαγή κάνουμε στο πεδίο εφαρμογή κινδυνεύει να επηρεάσει την χρηματοδότηση και την κατάσταση του ανταγωνισμού στην αγορά. Οπότε έχουμε κάποια ανησυχία. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να επικαιροποιηθεί το πεδίο εφαρμογή, αλλά φοβόμαστε τον πιθανό αντίκτυπο όσον αφορά και τον χρόνο υιοθέτησης του πακέτου που έχουμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Τιμπον, θέλατε να τοποθετηθείτε για τις ε, καθολικές αυτές υπηρεσίες. Θέλω να κάνω μία παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε. Με, υπό τη διεύθυνση του συναδέλφου Χάρμπορ πριν από την πρώτη ανάγνωση έγινε μια πολύ σημαντική εργασία η οποία ε, διεκπαιρεώθηκε σχετικά με αυτό το σχέδιο οδηγίας και κατέληξε σε συμβιβασμούς οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί και στην Επιτροπή και στη συνέχεια ή στην Ολομέλεια και που προσπαθούν να λάβουν υπόψη όλα τα εμπλεκόμενα συμφέροντα. Εγώ προσωπικά ε, θέλω το βασικό, δηλαδή η ουσία του ότι είχε ε, μπορέσει να γίνει αποδεκτό από τον Μάλκομ ε, ε, Harbour στην πρώτη ανάγνωση να μπορέσει να υιοθετηθεί σε δεύτερη ανάγνωση από την Ολομέλεια και να μην επιβαρύνουμε ε, ή να μην φορτώσουμε υπερβολικά ε, τον συμβιβασμό ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Αυτή την παρατήρηση θέλω να κάνω. Κύριε Χάρμπορτ, θέλετε να τα συνοψίσετε. Ναι ακούγοντας και αυτό το οποίο είπε ο Ζακ Τουμπον για τους συμβιβασμούς, δεν νομίζω πως είναι πολύ δύσκολο εμείς και η Προεδρία να καταλήξουμε σε ένα καλό κείμενο για τους καταναλωτές. Νομίζω ότι το πεδίο εφαρμογής ε, όσον αφορά αυτή τη στιγμή την παραβίαση των δεδομένων είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να αναζητήσουμε κάποια λύση αν και βεβαίω τώρα οι προσδοκίες μας είναι μειωμένε μετά από αυτά τα οποία μας είπε η Προεδρία αλλά θα ήθελα η Προεδρία να συναντηθεί μαζί μας, να μας αφιερώσει λίγο χρόνο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δηλαδή εγώ σέβομαι τους ηγητές, αλλά θα θέλαμε λίγο χρόνο, να μας αφιερώσουν λίγο χρόνο για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε στη δεύτερη ανάγνωση. Ναι, βεβαίως, λέει η πρόεδρο, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία γιατί είναι σημαντικό αυτό και για την Επιτροπή μας. Οπότε οπωσδήποτε σας στηρίζει η Επιτροπή μας και εσάς και τους ηγητές Νομίζω έχουμε προθεσμία για τις τροπολογίες μέχρι τις 11 Μαρτίου. Μέχρι τέλος Μαρτίου εξέταση των τροπολογιών και μετά θα έχουμε τον Απρίλιο ε, την ψηφοφορία. Κύριε Γκεπχάρτ, ναι, 11 Μαρτίου δεν έχω πρόβλημα, αλλά το κείμενο το έχω μόνο στα αγγλικά. Θα ήθελα να γνωρίζω πότε θα λάβω τη γερμανική μετάφραση. Δεν είμαι διατεθειμένη να αποδεχτώ, να εργαστώ μόνο με βάση το αγγλικό κείμενο. Με συγχωρείτε. Ναι. Να δω πότε θα είναι σε όλες τις γλώσσες διαθέσιμο. Νομίζω Δευτέρα 9 του μηνός. Οπότε η προθεσμία είναι 11. Ε, αν το κάνουμε πέμπτη, να δώσουμε τέσσερις μέρες, Μάλκομ, στους συναδέλφους, νομίζω είναι καλύτερο από δύο μέρες μόνο. Ελπίζω οι συνάδελφοι να μην καταθέσουν πολλές ε, τροπολογίες, γιατί κατά βάση είναι η θέση που έχουμε υιοθετήσει ήδη. Και ούτως ή άλλως έχουμε και συμβαστικές τροπολογίες με τους γεωδησίγητες, αλλά βεβαίως είναι δικαίωμα των συναδέλφων να καταθέσουν τροπολογίες, αλλά είναι αρκετά μεγάλη αυτή η δεύτερη ανάγνωση, λόγω του χρόνου βεβαίως και λόγω των διαπραγματεύσεων που δεν είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε με την Προεδρία. Ναι, πρέπει μέχρι 31 Μαρτίου όμως να ψηφίσουμε, γιατί τότε είναι η τελευταία συνεδρία. Οπότε κυρία Γκέπχαρτ θέλετε, μία εβδομάδα θα σας φτάσει. Ελπίζω. Ελπίζω να μην χρειαστεί να καταθέσω καμία τροπολογία, Μάλκομ. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι εδώ πέρα ένα πολύ σημαντικό η καθολική παροχή υπηρεσιών και θέλω να το δω με την ησυχία μου αναλυτικά στα γερμανικά για να μπορέσω να αξιολογήσω και να δουλέψω κιόλας. Οπότε Πράγματι θα ήθελα άλλες δύο μέρες γιατί γνωρίζω ότι δεν έχουμε μόνο αυτό το κείμενο αλλά και άλλα πράγματα που παράλληλα πρέπει να γίνουν. Okay, so, so can we... Λοιπόν, τότε αν συμφωνήσουμε θα δώσουμε μία επιπλέον ημέρα, θα έχουν τη Δευτέρα το ε, το κείμενο στη γλώσσα τους και μέχρι την Πέμπτη θα έχουν χρόνο να διατυπώσουν τροπολογίες, δηλαδή μεταφέρουμε ε, στις 12 του μηνός. Ε, τώρα θα ψηφίσουμε. Ελπίζω ότι όλοι είσαστε εδώ και να έχουμε τον κατάλογο όλων των ψηφοφοριών. Το πρώτο είναι η ομιλία, το κείμενο του κυρίου Καμάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι όσοι παρακολούθησαν τις τελευταίες συζητήσεις για τις τροπολογίες θα είδαν ότι δεν υπήρχε δυνατότητα συμβασμών και ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις συγητές όλων των ομάδων ε, και το προσωπικό τους γιατί νομίζω ότι ιδίω τα θέματα της διαφάνειας έχουμε καταλήξει σε καλούς συμβιβασμούς και ε, θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στην πρόταση Επιτροπής πολύ σύντομα. Θέλω όμως να ευχαριστήσω τους σκιώδεις και το προσωπικό τους για την εξαιρετική συνεργασία. Θαυμάσια συμφωνείτε βλέπω και κανείς άλλος δεν ζητά το λόγο θα ήθελα να ψηφίσετε είναι η πρώτη φορά που ψηφίζουμε έχετε τις ε, κάρτες σας είναι πρώτη φορά που ε, ψηφίζουμε εδώ και έτσι καλό είναι να έχετε τις κάρτες σας ώστε ηλεκτρονικά να μπορούμε να το ελέγξουμε έχετε όλοι μία ε, κάρτα ψηφοφορίας Ο κύριος μαντάς θα χρειαστεί να ψηφίσουμε με την, ε, με την κάρτα διότι είναι πιο γρήγορο ο χειρός. Ναι, αλλά σας είπα ότι θα πρέπει να σαρώνουμε κατά κάποιον τρόπο όλο το χώρο ε, εάν ε, είναι εύκολο θα το κάνουμε ε, δια ανατάσεως χειρός αλλά είδαμε είχαν πει στην προηγούμενη συνεδρία να φέρετε τις κάρτες σας δηλαδή όσοι δεν έχουν κάρτες θα πρέπει να φέρουν μία πέστε στη βοηθό σας παραδείγματος χάρη να φέρει μία το είχαμε ήδη ειδοποιήσει την προηγούμενη φορά δεν σας είπα ότι θα σας αποκλείσω. Είπα ότι θα αρχίσουμε να ψηφίζουμε διανατάσεως χειρός. Ζητήστε στο προσωπικό σας να σας φέρουν κάρτα και διαφορετικά θα πρέπει να σας, ψηφί, να σας μετρήσουμε χωριστά και καθυστερούμε. Το, η τροπολογία έξω κυρίου Καμάλ, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. τροπολογία 34, υπέρ. Τώρα πρέπει να μετρήσουμε. Κατά. Αποχές. 17 υπέρ, 10 κατά, χωρίς αποχές. Άρα εγκρίνεται. 35 καταπίπτει, πάμε στο 7 δέλτα, υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. Άρθρο 2, τροπολογία 8. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 9. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11 πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το 37 του κυρίου Κράμερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά και αποχές απορρίπτεται 13 ε, κατά 12 υπέρ ε, βλέπετε όμως γι' αυτό ζήτησα να έχετε τις κάρτες σας απορρίπτεται άρα τώρα παίρνουμε το 11 ο δεύτερο τμήμα του κυρίου Καμαλιπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Άρθρο 4. 11 ε, τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αποσύρονται. Η 41 αποσύρεται, η 40 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Το 11 τέταρτο τμήμα ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 του κυρίου Νιούτον Τάν υπέρ. Κατά Απορρίπτεται. 9 υπέρ, 15 κατά. 4. Άρθρο 4. Ε, τροπολογίες για διαγραφή 11, 46, 47 υιοθετείται. Το 48 αποσύρεται. Το 49 ποιο είναι υπέρ. Απορρίπτεται. 50 υπέρ. Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Λοιπόν, για σηκώστε τα χέρια σας. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα το 11 έκτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές πορύπτεται. Άρθρο 4. 11 ε, του Καμάλ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 51 του Νιου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, το 11.8 ε, του κυρίου Ικαμάλ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 11-9 ε, υπέρ κατά απορρίπτεται, 11-10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 του κυρίου Μάντερς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 Νιούτον τάν υπέρ κατά αψοχές απορρίπτεται 57 Νιούτον τάν υπέρ θα πρέπει να μετρήσουμε να κρατήσετε τα χέρια σας αρκετή ώρα ψηλά κατά απορρίπτεται. Το 58 αποσύρεται. 59 της κυριας Χάντσλικ Χάνσλικ. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11-11 του κυρίου Καμάλ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, το 11-12 του κυρίου Καμάλ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην ε, πρώτη συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οπότε όλα τα υπόλοιπα του άρθρου 6 καταπίπτουν και τώρα πηγαίνουμε στη σελίδα 13 σύμφωνα με τον κατάλογό μου ε, άρθρο 6 παράγραφος 4 Μηχανισμοί ε, διαφυγής. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται επίση. Εγκρίνεται. Και πάμε στο 114 του κυρίου Σουάμπ. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 117-118 Σαλδεμός και Μπουρφών υπέρ Ας μετρήσουμε. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά για να δούμε. εγκρίνεται σαφώς. Κατόν δεκάξι. 116 της κυρίας Κάριν Ρίς Γιώργεσον υπέρ εγκρίνεται 119 του κυρίου Τουμπό υπέρ Κρατήστε λοιπόν τα χέρια σας ψηλά, ώστε υπέρ, κατά, Γκρίνεται 14 υπέρ, 13 κατά. Χωρίς αποχές. 120 του κυρίου Μπουλφόν υπέρ, κατά. Νομίζω περίφθη. Απερίφθη. 121. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 14 ε, απορρίπτεται. 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 123 του κυρίου Μπουλφόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 άρθρο 11. 15 του κυρίου Καβάλ όπου οι φιλελεύθεροι ζητούν χωριστή ψηφοφορία ποιος είναι υπέρ του πρώτου μέρους. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 μάντερς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 16 του Καμάλ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 του κυρίου Χάρβου 127 του κυρίου Χάρβου απορρίπτεται Τώρα προχωράμε στη 17 μπουλφών. Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Ποιος είναι υπέρ, για ξανασηκώστε τα χέρια σας. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε τα εκτιμώντας 2 5, τροπολογία Νετ Καμάλ απορρίπτεται. Ένα δεύτερο μέρος απορρίπτεται επίσης, τροπολογία 18, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 19 του κυρίου Νιούτον Τάν υπέρ Κατά. 18. So 10 in favor, 18 against, that's clearly rejected. Απορρίπτεται. Ε, τροπολογία Αρμάντε, περ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1, τρίτο μέρος Καμάλ απορρίπτεται, 21 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, με συγχωρείτε, 15 υπέρ, 12 κατά. Τώρα έχουμε την ε, τροπολογία 1 τέταρτο μέρος του κυρίου Καμάλ. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1 πέμπτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22. Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί αυτό. Μετά ε, ε, ένα έξι καμάλ απορρίπτεται. Μετά έχουμε την 1-7 του Καμάλ και πάλι απορρίπτεται. 23 δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. 1-8 Ντέτ Καμάλ απορρίπτεται. 1-9 του Καμάλ επίσης απορρίπτεται. 24 δεν ψηφίζεται. 1-10 το τμήμα του Καμάλ απορρίπτεται. 2 Πρώτο μέρος του κυρίου Καμάλ απορρίπτεται. Αφού αυτός δεν τις υποστηρίζει, γιατί ψηφίζουμε αυτές τις τροπολογίες. Απορρίπτεται. 25. Απορρίπτεται επίσης. 2-3 του κυρίου Καμάλ. Απορρίπτεται. 26. Μπουλφόν υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται για να δούμε και πάλι 26 26 Κατά και μία αποχή. 15 υπέρ, 15 κατά απορρίπτεται. Γι' αυτό είναι πιο εύκολα αυτά να γίνεται με τις κάρτες. Το 27 δεν χρειάζεται να το ψηφίσουμε. Τροπολογία 3 καμάλ, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 δεν χρειάζεται να ψηφιστεί, 29 ούτε. 4D του κυρίου Καμάλ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 σβάμπ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 Βουλφόν υπέρ κατά αποχές Τροπολογία Καμάλ 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 της κυρίας ε, Κάριν Σιν Γιόγκεσεν πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ κατά νομίζω ότι εγκρίθηκε νομίζω εγκρίθηκε με 17 υπέρ 10 κατά και χωρίς αποχές οπότε δεν ψηφίζουμε την 33 και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του γνωμοδότησης ποιος είναι υπέρ παρακαλώ κρατήστε τα χέρια σας ψηλά Αποχές 18 υπέρ και 14 αποχές. Συγκαρητήρια κύριε Καμάλη. the results again, Madam Chairman. Αποτελέσματα, κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Okay, um, Ωραία. Θα συνεχίσουμε την επόμενη ψηφοφορία. Έχετε τον κατάλογο ψηφοφοριών μπροστά σα. Ή ε, αν ναι, έχετε τον κατάλογο. Πρώτα απ' όλα ποιος δεν έχει την κάρτα του. Κάρτα ψηφοφορίας. Την έχετε όλοι. Εντάξει. Θα πείτε κάθε φορά που το ψηφίσετε μετά θα θα μετράμε. Πού είναι η κυρία Βόλη, η συγγετρία. Πρώτα απ' όλα, έχει η συγγετρία το λόγο. Αν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο πριν αρχίσουμε την ψηφοφορία. Thank you very much, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω κάτι. Θα Πρέπει να ψηφίσουμε. Πρέπει να πω ότι υπήρχαν κάποιες εξελίξεις από την τελευταία φορά που συζητήθηκε το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας πήρε από τις νομικές υπηρεσίες του Συμβούλιο της Νομοδοτής που τίθενται τα ίδια θέματα που έθεσα και εγώ για την συμβατότητα της απαγόρευσης σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς. Δεν φαίνεται λοιπόν να υπάρχει καλύτερη εναλλακτική λύση από αυτήν η οποία θα αντικατοπτρίζει την νομική θέση. Πρέπει να πω ότι βεβαίως πολλοί έχουν αντίθετη άποψη για το ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο. Πιστεύω λοιπόν ότι ο καλύτερο τρόπο να λύσουμε το όλο πρόβλημα είναι να ψηφίσουμε και θα δούμε πώ θα περάσει το θέμα αυτό στην Ολομέλεια και ποιο θα είναι μετά το επόμενο βήμα. Ούτω ή άλλω θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφου που με βοήθησαν να προετοιμάσω όλη αυτή την διαδικασία ψηφοφοριών. Θέλετε το λόγο, παρακαλώ, σύντομα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι Έχεις απογε... Ναι, πρέπει να αναγνωρίσουμε πως ε, δεν πρόκειται για νομική αλλά για πολιτική μάχη. Η Κομισιόν ε, γνωρίζει πως ε, μια τέτοια απαγόρευση δεν είναι δυνατή, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει τώρα να βρούμε μια πολιτική λύση. Ευχαριστώ. Κύριε Μάντερς, δεν είστε σκιοδησίτης. Δεν θέλω να ξεκινήσει η συζήτηση. Ναι, υπάρχει ολική απαγόρευση στην Ολλανδία και στο Βέλγιο και δεν ε, υπήρξε κάποια προσβολή στον ΠΟΕ. Α, κοιτάξτε, ας μην μπούμε τώρα στην νομική συζήτηση. Το είπε η κυρία Γόλης, έχει βγει η νομική γνωμοδότηση του Συμβουλίου, έχουμε ζητήσει μία και στο Κοινοβούλιο. Μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τα νομικά ζητήματα. Αυτό το οποίο πρέπει να λάβετε σήμερα είναι μια πολιτική απόφαση, συνάδελφοι, και μετά θα δούμε. Ας... Ε, Αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία. Τροπολογία 1 της κυρίας Βόλης. Ψηφίζουμε. Δεν θα κάνουμε ηλεκτρονική ε, ψηφοφορία. Θα μετρήσουμε. Is everybody voted? Okay, close the vote. Αρχίζει η ψηφοφορία, λίγη ψηφοφορία. Ψήφισαν 30. 7 υπέρ, 22 κατά μία εποχή. 18 της κυρία Βόλης. Αρχίζει η ψηφοφορία. Καλύτερα να προχωρήσουμε έτσι η ψηφοφορία. 7 in favor, 23. 7 υπέρ, 24 κατά. Καμία εποχή. Απορρίπτεται. 82. Έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία. Ναι. Ναι. Πρώτα όλη την 82 ε, και μετά την, χωριστά τη λέξη ναν. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Όλη την 82. Υπέρ. Ε, συγγνώμη, αρχίζει η ψηφοφορία. 23 υπέρ, 24 υπέρ, 7 κατά. Δεν χρειάζεται να σας τα λέω, τα βλέπετε τα αποτελέσματα στην οθόνη. Τώρα, ψηφίζουμε χωριστά τη λέξη «ναν» για να την διαγράψουμε. Λοιπόν, τώρα για την ε, διαγραφή της λέξης none. Για διευκρινίστε, τι ακριβώς ζητάτε. Εγκρίθηκε η τροπολογία 82, έτσι. Τι ακριβώς θέλετε. Εντάξτε, για να σας πω ποια είναι η πρότασή μου. Εγκρίθηκε ολόκληρη η 82 και τώρα θέλω εγώ να φύγει η λέξη νον. Αυτό προτείνω να ψηφίσουμε. Να φύγει η λέξη νον. Εντάξει, κατάλαβα. Ακούστε, ψηφίσαμε με το non-commercial exchange, τώρα θέλετε το non να διαγραφεί. Εντάξει. Εάν είστε υπέρ της διαγραφής του νον... Ελπίζω να το καταλάβαμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Υπέρ λοιπόν αν θέλετε να διαγραφεί η λέξη non από το commercial exchange. Να είναι μόνο commercial exchange, όχι non-commercial exchanges. Okay. Okay, anyway, we have a result, so... <laughs> 21 υπέρ λοιπόν, 9 κατά, 22 υπέρ. Καμία εποχή. Άρθρο 2, τροπολογία 84. Υπέρ. Μάλλον ας αρχίσει ψηφοφορία. Τροπολογία 84. Λίγη ψηφοφορία. 25 υπέρ 6, καμία εποχή. Τροπολογία 86. Αρχίζει η ψηφοφορία. «29 υπέρ, 2 κατά. Εγκρίνεται». Άγκρη 13. Αρχίζει ψηφοφορία. Θέλετε κάποιες να τις ψηφίσουμε διανάταση των χειρών. Θα, της χειρός θα είναι πιο γρήγορο. Λοιπόν, άγκρη Λοιπόν, 13. Υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Ακούστε, κάποιες από αυτές θα τις ψηφίσουμε διανατάσεις της χειρός διότι ξέρουμε ότι είναι απολύτω σαφή τα αποτελέσματα. Θα πάμε πιο γρήγορα. Λοιπόν, 19 της κυρία Wallis. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 Wallis, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14 Άγκρι, υπέρ, Ηλεκτρονική ψηφοφορία στην Άγκρη 14. «22 προς 9. Εγκρίνεται. 88. σαλτεμόζε, Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 21 D κυρία Wallis. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 89 και NV16, 22 της κυρίας Βόλης, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 23 Βόλης, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στο άρθρο 2 Έχουμε ένα μπλοκ 24, 90, 90, 93, MV17 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνονται. Προφορική τροπολογία της Χαϊντιρούρου και Κρίστερ Σαλτεμόζε, 94, υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. 94, 18, 16 επρίπτονται. Προφορική 35 εγκρίνεται. Άρθρο 3. 25 Wallis στο άρθρο 3 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για τις απαγορεύσεις στο άρθρο 3. 25. Σαφές το αποτέλεσμα. 23 κατά απορρίπτεται. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε την επόμενη, δεδομένου ότι υπερψηφίστηκε η 96, αλλά ας ψηφίσουμε την 101 του κυρίου Μάντερς πρώτα απ' όλα. εάν η ενοποιημένη τροπολογία, εάν ε, προσθέσουμε εδώ τον όρο small scale, μπορώ εγώ αν θέλετε να αποσύρω την δική μου και να υποστηρίξω την ενοποιημένη. Ε, αν η κυρία Ρούλε και η κυρία Σάλντερ Μόζ ε, συμφωνήσουν, έχει καλώς. Ενοποιημένη τροπολογία λοιπόν ένα εγκρίνεται. Τροπολογία 102 άρθρο 3 παράγραφο 3 του κυρίου Μάντερς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 και 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται άρθρο 4 Ποιος είπε ότι θέλει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Θέλετε στην 103 και στην 104 ηλεκτρονική επαλήθευση. Έχει καλός. 103-104 λοιπόν. Αρχίζει η ψηφοφορία. 3 υπέρ 29 κατά. Ψαφέστατα τα πράγματα. Άρθρο 4. Ομάδα τροπολογιών 106, 105, 107, 108, NV 21. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 106 όχι 110 άρθρο 5 Πάλι έχουμε μία ομάδα τροπολογιών, 17, 18, 19, 23, υπέρ, κατά, καταπίπτουν Άρθρο 6, ομάδα πάλι τροπολογιών στο άρθρο 6, εγκρίνονται. Άρθρο 7, 39, 121, 122, 123, 24, υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Άρθρο 8, 124, 125, nv 25, υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Άρθρο 9, 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 126 ρούλε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 11 φορές 127, 128, 27, 28 της ΕΜΒΗ εγκρίνονται. Άγκρι δεν ψηφίζουμε τις άλλες. Τόν 29 και άγκρι 25 υπέρ. Τι κάνετε, δεν σηκώνετε το χέρι. Πρόκειται για προσθήκη. Ας κάνουμε. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, μπορώ να πω ότι είστε υπέρ αυτής της προσθήκης. Αποφασίστε να ψηφίσετε. Είμαστε λοιπόν υπέρ. 130. Έμπνερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 12. Άγκρι 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 40 Wallis υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 131-132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Δεν ψηφίζουμε την 27. Παράρτημα 1, 133, 134, NV29, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται, 135 καταπίπτει, παράρτημα 2, 137, 138, NV30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Όλες οι υπόλοιπες καταπίπτουν. Αιτιολογική σκέψη. Ε, μία καινούρια. Μπορούμε να την ψηφίσουμε. Υπάρχουν κάποιες μικρές γλωσσικές διαφορές ανάλογα με τις γλώσσες. Ε, NV4 εγκρίνεται, άγκρι 2 ως προσθήκη εγκρίνεται, άγκρι 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 447, ηλεκτρονική επαλήθευση. Οκτώ υπέρ 24 κατά απορρίπτεται. Άγκρι 3. Ε, συγγνώμη, ε, τη λογική σκέψη 3, άγκρι 5. Απορρίπτεται. 48-49, NV5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 ρούλε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 Wallis υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 ρούλε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 Wallis υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 ρούλε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 όχι Προφορική τροπολογία 53. Σάλμος Γούλε. Την έχετε μπροστά σα το κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση. Στην προφορική 53. Ωραία. Yeah, that's very clearly adopted. 23. Εγκρίνεται. 23 προς 9. 7 Wallis υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 8 Wallis υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 55 εντάξει ρούλε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Αιτιολογική σκέψη 11, 56, 57, 58, 59, ένβη 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συγγνώμη, η NV6 πρέπει να ψηφιστεί, όχι, ναι, πρέπει να ψηφιστεί ως προσθήκη η NV6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 καινούριο, 60, Held, Σαλτεμόζ, and Westlund, υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Άγριο 8, υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Εταιρική σκέψη 12, 62, 63, 64, NV9, υπέρ, κατά, εγκρίνονται. Τροπολογία 14 τελική σκέψη 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. με Μοτιμένη κοινή τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70. Η κυρία Βόλης υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 76. Όχι. Ναι. 76 έμπνερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13β71 του κυρίου Κρέμερ. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση στην 71 Κρέμερ. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά σκάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. 22 προς 10 εγκρίθηκε. Αιτιολογίες του 14, 14 MV11 υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται. Οι άλλε καταπίπτουν 16 τροπολογίες 77-78 MV12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. «81 Έμπνερ στην εταιρική σκέψη 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται». 17 Wallis υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεν ψηφίζουμε τη citation. Ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεσης στο σύνολό του έτσι όπως τροπολογήθηκε η ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει η Έλειξε ψηφοφορία. Η έκθεση λοιπόν έτσι όπως τροπολογήθηκε εγκρίνεται με 25 υπέρ 7 κατά και καμία αποχή. Διαδικαστικό κυρία Ματιού. Ευχαριστώ. Μπορείτε παρακαλώ να σημειώσετε ότι εγώ εξέφραζα τη θέση της μειοψηφίας στην έκθεση αυτή.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 Όχι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, συνάδελφοι, όσοι θα μείνουν για την ακρόαση και την κυρία Επίτροπο, καθίστε, οι υπόλοιποι παρακαλώ αποχωρήστε ήσυχα. Okay, thank you. Thank you very much. Sorry, we, sorry, we have a, uh, we had quite um, colleagues, could I ask you... Λοιπόν, συνάδελφοι, παρακαλώ αν θέλετε να συζητήσετε περάστε έξω γιατί έχουμε καθυστερήσει και 20 λεπτά. Ευχαριστώ. και θέλουμε να συνεχίσουμε με την ακρόαση για να μην χάσουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες που έχουν ταξιδέψει για να έρθουν εδώ. Οπότε εγώ δεν θα κάνω εισαγωγικά σχόλια γιατί έχουμε καθυστερήσει ήδη 20 λεπτά και θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Επίτροπο να μας πει λίγα λόγια για να κάνει μια εισαγωγή στην ακρόαση και μετά θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες μας γρήγορα και μετά θα έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις. Καλώς ήρθατε λοιπόν κύριε Επίτροπε, Είστε ευπρόσδεκτοι όπως πάντα και χαιρόμαστε που θα έχουμε σήμερα αυτή την σημαντική ανταλλαγή απόψεων που ελπίζουμε ότι θα συνεισφέρει στην τελική πρόταση για την οδηγία δικαιωμάτων των καταναλωτών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Χαίρομαι που έχω ξανά την δυνατότητα να μιλήσουμε για το πολύ σημαντικό ζήτημα των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Συγχαίρω την κυρία Μακάρθη, του συντονιστές και τη γραμματεία της Επιτροπής για το ότι οργάνωσαν αυτή την πολύ σημαντική ακρόαση την κατάλληλη στιγμή. Με στιγμή στις ε, συζητήσεις αντιλήφθηκα πως χρειάζεται πράγματι χρόνος. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο κείμενο. Η οδηγία θα διαμορφώσει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων καταναλωτών για τις επόμενες γενιές. Στόχος μου λοιπόν είναι να έχουμε καλύτερες τιμές και καλύτερη επιλογή για τους καταναλωτές και τα νοικοκυριά, να έχουμε δηλαδή σύγχρονα δικαιώματα για τους καταναλωτές και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Σε δύσκολους οικονομικούς καιρούς χρειαζόμαστε υγιείς αγορές με σωστούς κανόνες. Στους τελευταίους πέντε μήνες έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτή η οδηγία δικαιωμάτων των καταναλωτών και εγώ παρακολούθησα αυτή τη συζήτηση με πολύ προσοχή. Δεν πρόκειται εδώ πέρα για κάποιο κάποια επιλογή μεταξύ υψηλού επίπεδου προστασίας των καταναλωτών και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θέλουμε και να προστατεύσουμε τους ε, καταναλωτές ε, οπωσδήποτε, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να έχουμε κατά νου και τα πραγματικά πλεονεκτήματα που μπορεί να φέρει η εσωτερική αγορά σε κάθε νοικοκυριό. Για όσου θεωρούν πως δεν έχουν σημασία οι τιμές για τους καταναλωτές, πρέπει να το ξανασκεφτούν. Όσοι θεωρούν ότι η μεγαλύτερη επιλογή είναι κάτι προαιρετικό, πρέπει και αυτοί να το ξανασκεφτούν. Όσοι επίσης θεωρούν πως η εσωτερική αγορά είναι μια πολυτέλεια σε μια εποχή κρίσης και αυτοί πρέπει να το ξανασκεφτούν. Αυτή η οδηγία δεν ε, εμποδίζει τα κράτη-μέλη από το να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της οδηγία και για συναλλαγές μέσω, ε, μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Έχουν την δυνατότητα τα κράτη-μέλη να ρυθμίσουν εκείνες τις πτυχές που είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής οδηγίας. Η οδηγία αυτή επίσης δεν αποτρέπει τα κρατη από το να απαγορεύσουν τα τηλεφωνήματα τα οποία δεν έχει ζητήσει κανείς. Μπορούν αυτό να το επιβάλλουν τα κρατημέλη με οποιοδήποτε μέσο, είτε πρόκειται για πρόστιμα είτε πρόκειται για την ακυρότητα της σύμβασης. Δεν εξαναγκάζει επίσης αυτή η οδηγία τα κράτη-μέλη να μην έχουν την δυνατότητα απόρριψη παραδείγματο χάρη ελαττωματικών αγαθών ή οποιαδήποτε άλλη εγγύηση που παρέχει το συμβατικό τους δίκαιο, όπως παραδείγματο χάρη στη Γαλλία στο Βέλγιο. Αυτό, αυτή η οδηγία επίσης δεν υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να μην εφαρμόζουν πλέον τις νομικές τους εγγυήσεις σε υπηρεσίες όπως παραδείγματο χάρη κατασκευές ή ψηφιακές υπηρεσίες. Ε, λυπούμε για το ότι οι συζητήσεις πρόσφατα φαίνεται πως αγνοούν το ότι υπάρχουν ουσιαστικά νέα δικαιώματα καθώς και ενίσχυση των υπαρχόντων δικαιωμάτων για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα έχουν τα δικαιώματά τους να βελτιώνονται, θα έχουν περισσότερα δικαιώματα με την παραλαβή και θα υπάρχει πράγματι προστασία για τυχόν ζημία των αγαθών μέχρι την πλήρη παραλαβή τους και θα υπάρχει και προστασία σε περίπτωση υπάρχουν κάποιες κρυφές χρεώσεις. Δεν θα χρειάζεται κάτι τέτοιο. Επίσης υπάρχει μία περίοδος υπαναχώρηση 40 ημερών. Για πρώτη φορά επίσης υπάρχει πανευρωπαϊκή απαγόρευση στο να συμπληρώνει κανείς εκ των προτέρων ε, κουτάκια. Επίσης θα υπάρχει επέκταση της εγγύησης ανεξαρτήτως της αξίας της συναλλαγής. Επίσης θα μπορούν να υπαναχωρήσουν είτε με ένα χειρόγραφο γράμμα είτε με ένα απλό email οι καταναλωτές. Επίσης θα υπάρχει υποχρέωση στις συμβάσεις στο διαδίκτυο, π.χ. στο eBay, θα πρέπει να αποκαλύπτει κανείς ότι είναι έμπορος και όχι καταναλωτής. Επιπλέον, χάρη στα νέα ενιαία ευρωπαϊκά δικαιώματα θα μπορούμε να έχουμε μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης για τα δικαιώματα κατά τη στιγμή της πώληση, κάτι παρόμοιο με αυτό το οποίο υπάρχει για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών εταιριών. Πολύ σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα για μένα και ελπίζω να έχω την υποστήριξή σας. Ακούστηκαν κάποιες ανησυχίες για το πεδίο αυτής της πρότασης, παραδείγματος χάρη για το ψηφιακό περιεχόμενο. Γνωρίζετε πως έχω δεσμευτεί για να βελτιωθεί η προστασία των καταναλωτών ψηφιακών προϊόντων και εργάζομαι σκληρά. Αλλά γεγονό είναι πως ε, χρειαζόμασταν περισσότερο χρόνο για να βρούμε τα προβλήματα στον τομέα αυτών και υπόσχομαι να επανέλθω σε αυτό το ζήτημα του ερχόμενου μήνε. Ως Ερετή εκπρόσωποι των πολιτών εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζετε καλύτερα τι ανάγκε των καταναλωτών όπου και αν ζουν και ψωνίζουν. Έχοντα συναντηθεί με πολλούς από εσά, με οργανώσεις καταναλωτών, με εμπειρογνώμονες, με τις εθνικές αρχές, αναγνωρίζω πως σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν θεμητές και κατανοητές ανησυχίες για κρίσιμα ζητήματα. και θεωρώ ότι τα εξής είναι τα σοβαρότερα. Εάν η διετής εγγύηση επαρκεί εάν το βάρος της αποδείξεως ε, και η εξάμεινη περίοδος εντός της εγγύησης είναι ε, δίκαιο για τους καταναλωτές. Εάν ο τρόπος ε, της επανόρθωσης ο οποίος προτείνεται είναι σωστό, Μήπως θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότεροι όροι συμβάσεων στη μαύρη λίστα του παραρτήματος. Συμφωνώ να δούμε αυτά τα ζητήματα. Ίσως κάποια δικαιώματα των καναλτών πρέπει να ενισχυθούν. Η οδηγία αυτή τη στιγμή είναι πλέον στα δικά σας χέρια και είμαι σίγουρη πως ε, θα βρείτε την σωστή ισορροπία για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών αλλά και για να έχουν και οι επιχειρήσεις λειτουργικούς κανόνες. Αλλά δεν είμαι διατεθειμένη να συμβιβαστώ στην αρχή του να έχουμε ενιαίους κανόνες που θα ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις και όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές από το μαγαζί που έχουν απέναντί τους στη γειτονιά μέχρι ε, το διαδίκτυο. Τώρα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε αγορές που θα λειτουργούν αποτελεσματικά, που θα δώσουν στις επιχείρησεις την σταθερότητα που χρειάζονται και εμείς χρειαζόμαστε από αυτές, αγορές οι οποίες θα επιτρέψουν στους καταναλωτές να αγοράζουν τα αγαθά που χρειάζονται, όπου και όποτε τα χρειάζονται, στη σωστή τιμή. Όλοι μας στην περίοδο αυτή της οικονομικής κρίσης οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού και να συνεισφέρουμε στην ανάκαμψη. Οπότε μια υγιής αγορά χρειάζεται δυνατούς κανόνες όσον αφορά την επιβολή και βεβαίω και κανόνες επανόρθωσης, κάτι το οποίο θα γίνει με εναρμονισμένους κανόνες. Όσοι από εμά είμαστε αρκετά τυχεροί να έχουμε θέσεις εργασίας, μειώνουμε τις δαπάνες μας. Όσοι έχασαν τη δουλειά τους αναγκάζονται να κάνουν ακόμη περισσότερες μειώσεις. Οπότε, εάν υπήρχε κάποια στιγμή στην οποία χρειάζονταν διαβεβαίωση για το τι αγοράζουν οι καταναλωτές και για το ότι θα έρθει την κατάλληλη στιγμή και είναι αυτό το οποίο χρειάζονται, η στιγμή αυτή είναι τώρα και τώρα πρέπει ο Ευρωπαίος νομοθέτης να δώσει αυτή τη διαβεβαίωση. Η ιστορία μας διδάσκει πως εάν αν όλοι τα παρατήσουμε και μείνουμε σπίτι μας και δεν αγοράζουμε τίποτα και δεν πουλάμε τίποτα θα είναι χειρότερη και πιο μακροπρόθεσμη η ύφεση. Αλλιώς θα χρεοκοπήσει η Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να έχουμε την δυνατότητα να δημιουργηθούν αυτές οι εμπορικές ροές δισεκατομμυρίων ευρώ σε ολόκληρη την Ευρώπη που θα δημιουργήσουν και αυτές ε, σε δημιουργία θέσεων εργασίας. Ελπίζω να με γνωρίζετε. Πια έχω ακούσει και θα ακούσω τις ανησυχίες σας, θα σημειώσω και την κριτική που θα ασκήσετε και ελπίζω όλοι να δείτε με ανοιχτό μυαλό και με ευρωπαϊκή νοοτροπία αυτή την πρόταση και σας βεβαιώ πως η Κομισιόν επίσης θα είναι ανοιχτή να ακούσει επικοδομητικά σχολεία, αν βασίζονται σε στοιχεία. Είμαι πεπισμένη πως ενιαίοι κανόνες και υψηλό επίπεδο προστασία συμβαδίζουν. Είμαι επίσης πεπισμένη πως τις ε, διαπραγματεύσεις το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα βρουν τη σωστή ισορροπία για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες μας και καταναλωτές στον 21ο αιώνα. Έχω ξεκαθαρίσει επίσης πως ε, είμαι διατεθειμένη να μείνω εδώ μαζί σας μέχρι το τέλος ε, της ακρόασης και χαίρομαι που με φιλοξενείτε. Θα ακούσω τις ανησυχίες σας και εύχομαι να έχουμε καλή δουλειά και καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you, So I think you... Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Νομίζω ότι τώρα έχετε ε, οριοθετήσει το θέμα. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω τώρα γιατί θα ήθελα να αφήσω το χρόνο στους εμπειρογνώμονες και για να καλύψουμε την καθυστέρηση. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στην πρώτη συνεδρίαση που έχει σαν ε, επικεφαλίδα οι εμπειρίες αγοραπολισιών διασυνοριακά, ε, η εναρμόνιση της, του προτινόμενου πλαισίου νομοθεσίας καταναλωτών. Η ε, Γιούτα Γκάρκμαν είναι η οποία θα μιλήσει από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών το οποίο στηρίζουμε. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω για την διασυνοριακή εργασία των καταναλωτών. Ε, πάρα, πολλά, πάρα πολύ σύντομα θέλω να σας μιλήσω για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτού. Ε, φαντάζομαι το γνωρίζετε αλλά για όσους το αγνοούν θα ήθελα να διευκρινίσω. Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών είναι ε, ένα δίκτυο που έχει καταρτιστεί το 2005 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει σαν στόχο να στηρίζει τον ε, καταναλωτή σε θέματα διαφορών ε, και να συμβάλλει σε εξοδικαστικές ε, ε, ρυθμίσεις. Υπάρχουν διάφορα κείμενα, κέντρα στην Ισλανδία, στην Νορβηγία και το κέντρο στο ΚΕΛ το οποίο συνδυάζει το κέντρο για τη Γαλλία και για τη Γερμανία καθότι βρίσκεται στα σύνορα των δύο χωρών. Έχω φέρει και ορισμένους αριθμούς μαζί το 2007 ε, το είχαμε δεχθεί ε, 22.000 ερωτήσεις ε, και 29.000 ε, ε, ερωτήματα εκ των οποίων μεταφράσαμε και διεκπαιρεώσαμε 20.000 περιπτώσεις διαφορών και ιδίως επικεντρωθήκαμε σε ρυθμίσεις εξοδικαστικές. Δηλαδή τα κέντρα αυτά προσπαθούν να βρουν εξοδικαστικά μία ρύθμιση για έναν τομέα όπου επιτυχάνουν μάλιστα σε ένα μεγάλο ποσοστό. Την επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Δύο τρίτα των περιπτώσεων τα οποία έχει διεκπαιρεώσει το Γερμανικό Κέντρο είναι συμφωνίες για, ε, εμπόριο στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ αλλά α, αντιστοίχως 29% είναι περιπτώσεις συναλλαγών εις το κατάστημα και ένα ποσοστό είναι συναλλαγές ε, ε, από πλασιέ πόρτα-πόρτα. Ως επιτοπλίστων αναφερόμαστε σε ε, ρήτρε συμφωνιών και στις παραδόσεις όπου είτε η παράδοση δεν είναι σωστή δεν υπάρχει καθόλου παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων και ε, κοιτάμε και επίσης περιπτώσεις εγγύσεως. Δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένους αριθμούς αλλά υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες ε, ε, οφείλονται σε διαφορετική νομοθετική κατάσταση στα δύο κράτη. Δηλαδή ένα προσωστό το οποίο επίσης δεν μπορώ να προσδιορίσω και πρέπει να αξιολογηθεί αναφέρονται σε διαφορετικό δίκαιο καταναλωτών και επίσης ε, για τελείως ε, διαφορετικό ε, ενοχικό δίκαιο. Επίσης υπάρχουν δικαιώματα όπου έχει παραβιαστεί το δίκαιο και επίσης περιπτώσεις όπου η επιχείρηση δεν τα δικαιώματα του καταναλωτή. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ε, προσφέρει να ε, ταξινομήσουμε τις περιπτώσεις μας αναλόγως των αποτελεσμάτων. Βασικά όμως θέλω να αναφερθώ εδώ σε τρία σημεία, διότι για τους καταναλωτές το πρόβλημα το οποίο ε, δημιουργείται είναι ότι πολλοί δεν θέλουν να δώσουν τα εμπορεύματα διασυνοριακά και αυτό οφείλεται σε διαφορετικές σημάνσεις, σε διαφορετική πληροφόρηση και ε, ε, είναι ε, επίσης περιπτώσεις άρνησης μιας μεγάλης επιχειρήσεως να παραδώσει τα υλικά σε μια άλλη, τα εμπορεύματα σε μια άλλη χώρα. Υπάρχουν επιπλέον και καταναλωτές οι οποίοι κατά την πείρα μας δεν γνωρίζουν καν το εθνικό τους δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ε, έχει σημειώσει τον ε, νομικό κατακερατισμό, ο οποίος υπάρχει και ο οποίος πρέπει να επιληθεί διότι οι καταναλωτές ξέρουν ε, σχετικά λίγο ποια είναι τα δικαιώματά τους στη χώρα τους ξέρουν ότι υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιο δίκαιο ξέρουν επίσης ότι ε, μπορούν να έχουν προσφυγή σε περίπτωση που κάνουν διασυνοριακές ε, αγορές αλλά ε, ε, ε, για μας το σημαντικό είναι η άρνηση της διασυνοριακής πώληση και επίσης υπάρχουν και ορισμένες εταιρείες όπου βλέπουμε ότι ορισμένες χώρες έχουν, ε, ε, ε, έχουν θηγατρικές εταιρείες παραδείγματος χάρη στη Γαλλία όπου όλοι οι κωδικοί των προϊόντων είναι τα ίδια αλλά πέραν αυτού δεν ε, ε, είναι ίδιες οι τιμές και για, λόγω των διαφορών των τιμών δημιουργούνται προβλήματα. Υπάρχουν όμως πολύ πιο σοβαρά προβλήματα με τις μικρομεσαίες επιτυχηρήσεις και αυτό διότι ουσιαστικά δεν γνωρίζουν ποιο είναι το δίκαιο που διέπει την άλλη χώρα, ποια είναι τα δικαιώματα και εκεί έχουμε πολλά προβλήματα. Ε, οι λόγοι για τους οποίους δημιουργείται κάτι τέτοιο και πρέπει να υποφεληθούν οι καταναλωτές από την εσωτερική αγορά ε, είναι θέματα επιβολής του δικαίου και Πολλές φορές οι καταναλωτές ε, προτιμούν να συναλλάσσονται με εμπόρους τους οποίους γνωρίζουν, που έχουν αποδειχτεί σοβαροί και επίσης ένα πολύ βασικό θέμα είναι ε, η δυνατότητα ή έλλειψη συνεννοήσεως λόγω της γλώσσας. στην ε, την Γερμανία υπάρχει η δυνατότητα να στηρίξει κανείς το εσωτερικό εμπόριο και αν υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις από την ε, πείρα μας διαπιστώνουμε ότι ο λόγος για τους δισταγμούς για την εσωτερική αγορά είναι, ε, οφείλεται στην διαφοροποίηση των τιμών αναλόγως των χωρών ε, και οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν την αγορά για λόγους κόστους στις διάφορες χώρες και δεν έχουν μια σφαιρική εικόνα όσον αφορά την, ε, το σχέδιο της οδηγίας εγώ θα είχα να πω ότι μία συγκεκριμένη εναρμόνιση και εδώ θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ε, θέλει να δημιουργήσει, θέλησε να δημιουργήσει ένα δίκτυο ε, νομίζω ότι αυτό θα βοηθούσε ε, τις διασυνοριακές συναλλαγές και ιδίως όσον αφορά τη νομική βεβαιότητα διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ασάφεια υπάρχουν δηλαδή διαφορετικοί ορισμοί και όροι Υπάρχουν ε, ο καθορισμός και ο υπολογισμός των προθεσμιών η ε, ε, ανασφάλεια σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο και τέλος η ερμηνεία των εθνικών δικαστηρίων τα οποία ερμηνεύουν διαφορετικά τα δικαιώματα. Επίσης δεν θέλουμε να υπάρξει μία μείωση της προστασίας του καταναλωτού. Σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να κοιτάξουμε όλους τους κανόνες και να δούμε εάν πρέπει να παραμείνουμε σε μία ελάχιστη εναρμόνιση ή να έχουμε μία μια πλήρη εναρμόνιση σε υψηλό επίπεδο διότι μία μείωση της προστασίας του καταναλωτή η οποία αναφέρεται κατά καιρού, κατά τη γνώμη μας θα τάραζε την εμπιστοσύνη των ε, καταναλωτών και από την εργασία μας ιδίως ε, εφέτος ε, πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές είδαμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να ευαισθητοποιήσουμε τον καταναλωτή τον πολίτη να του δώσουμε μια θετική εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εφόσον ε, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προσέχει πολλά θέματα όπως είναι τα δικαιώματα του καταναλωτού και την προστασία του την οποία μπορεί κανείς να βελτιώσει σε πολύ ψηλό βαθμό και <clears throat> έτσι έχει αυξηθεί και η προστασία σε πολλές χώρες πράγμα το οποίο ε, καθημερινά ε, έχει ε, αισθητές επιρροές στους καταναλωτές. Το μήνυμα λοιπόν το οποίο μπορεί κανείς να δώσει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφεύγει να μειωθεί η προστασία του καταναλωτού σε εθνικό επίπεδο και επίσης αν δοθεί το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εναρμονίζει την προστασία των καταναλωτών σε ίσο επίπεδο σε όλες τις χώρες θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί διότι οι καταναλωτές πρέπει να το κατανοήσουν σωστά. Δηλαδή οι καταναλωτές δεν διαχωρίζουν το γενικό ενοχικό δίκαιο και το δίκαιο των καταναλωτών. Αν τους πούμε λοιπόν ότι έχετε τα ίδια δικαιώματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργείται ε, μία διαφορά διότι ε, είναι ε, έννοιες που δεν μπορούν να εξηγηθούν στον καταναλωτή και αυτά οδηγούν σε μεγάλη απογοήτευσή του πράγμα που είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ε, προσέξει κανείς πάρα πολύ, να το σταθμίσει, να κοιτάξει, να προωθήσει τα προσόντα της εσωτερικής αγοράς που είναι προς όφελος του καταναλωτή, διότι κατά τη γνώμη μου, εάν κοιτάξουμε κανόνα προς κανόνα την έκταση της ε, πλήρους εναρμονήσεως και ε, ποια ποιες νομοθεσίες επιτρέπουν στον καταναλωτή να χρησιμοποιήσει την εσωτερική αγορά θα ήταν ένα πολύ βασικό θέμα και θα μπορούσε να ρυθμιστεί και θα υπήρχε ένα σύστημα στο οποίο όλοι θα μπορούν να επαφίενται και όπου οι καταναλωτές θα μπορέσουν να υποφεληθούν από την εργασία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στον τομέα του δικαιωμάτων καταναλωτή. Ευχαριστώ. Σας δίνω λίγο περιθώριο, αλλά δεν θέλω να μακρηγορήσετε πάρα πολύ. Περνάμε στον κύριο Κάρλος Αλμάρης από την Business Europe που θα αναφερθεί στα πρακτικά προβλήματα για τις επιχειρήσεις της διασυνοριακές συναλλαγές και αν μπορούν αυτά να ξεπεραστούν από την πρόταση της Κομισιού. Δεν θα διαβάσω τα, τα βιογραφικά σας γιατί είναι και μακροσκελή. Γιατί είναι Όλοι εξαίρετε εδώ πέρα οι εμπειρογνώμονες μας. Απλά παρουσιάζω τους ε, εμπειρογνώμονες. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Σάλβαρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και την κυρία Μακάθη που κάλεσε την Business Europe να σας παρουσιάσει κάποιες απόψεις. Θα ασχοληθώ με τρία θέματα. Πρώτα απ' όλα να σας εξηγήσω πώς η business community πιστεύει ότι πρέπει να αναλυφθεί δράση στον τομέα αυτό. Δεύτερον, θα ήθελα να τονίσω πόσο επικοδημητικό είναι να γίνει μια θετική συζήτηση και τρίτον θα αναφερθώ στο περιεχόμενο της πρότασης. Κανένας ε, δεν θέτει σε αφισβήτηση το ότι λειτουργεί σωστά η ενιαία εσωτερική αγορά. Υπάρχουν κάποια διασυνοριακά θέματα, η διαδικαστικά, διοικητικά, προσωπική επιλογή. Η μεγάλη ποικιλομορφία που υπάρχει σε σχέση με αυτούς τους τομείς σε εθνικό επίπεδο πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα για την ε, ελεύθερη ε, διακίνηση αγαθών μεταξύ άλλων. Υπάρχουν λοιπόν αμοιβέ υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που κάνουν πωλήσει ε, διασυνοριακών και θα πρέπει να σέβονται όλες τις υποχρεώσεις τους. Υπάρχουν βεβαίως ε, κάποιοι κανόνες που ισχύουν εξαιτία ε, της ε, εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου και δημιουργούν κάποια προβλήματα. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το, ο κόστος συμμόρφωσης για να μπορέσει κανείς να συμμορφωθεί στην κοινοτική νομοθεσία είναι υψηλότερο. Υπάρχουν και άλλα θέματα όπως Μα εξήγησε και η προηγούμενη ομιλήτρια. Οι διάφορες ερετίες, κυρίως οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρές, πολλές φορές δεν μπορούν ε, να ασχοληθούν με τέτοιου είδου εμπόριο ή έχουν και ενδιασμού να το κάνουν, αλλά και οι καταναλωτέ χάνουν από αυτή την κατάσταση, ιδιαίτερω διότι έχουν λιγότερη επιλογή και δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αγαθά των άλλων κρατών μελά. Η αβεβαιότητα λοιπόν και η δυσπιστία στην αγορά εξαιτία ε, τη διαφορετικού επίπεδου προσήλωση των κρατών είναι κάποιο το αρνητικό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι και η οικονομία και η ενιαία εσωτερική αγορά χάνει αυτό το θέμα. Η οδηγία της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών θέλει να εφαρμόσει την καλύτερη δυνατή νομοθεσία του κανονισμού και η πρόταση έχει στόχο να το κάνει αυτό με την μίεση κάποιων ε, διαφορών που υπάρχουν ε, στα διάφορα δίκαια και θέλει συγχρόνως να αυξήσει την προστασία των κανατών. Για την Business Europe και τις ε, διάφορες ομοσπονδίες τις οποίες εκπροσωπούμε είναι σαφές τι πρέπει να γίνει. Πιστεύουμε λοιπόν ότι σωστά εμείς είμαστε υπέρ της εναρμόνισης, υπέρ της οδηγίας ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε καλύτερα τους στόχους που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά αναγνωρίζουμε ότι η συζήτηση δεν είναι απολύτως σαφής, διότι η... από τη μια υπάρχει η ποικιλία κανόνων και από την άλλη η τάση εναρμόνισης. Πιστεύουμε όμως ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει και είναι απαραίτητη κυρίως στα πλαίσια της μεγάλης οικονομικής κρίσης στην οποία διερχόμεθα σήμερα. Πριν να μπω στις λεπτομέρειες της πρότασης, θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια συζήτηση καλά δομημένη μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι κυρίως σε εθνικό επίπεδο η πρόταση εξετάζεται αποκλειστικά από την ε, εθνική οπτική γωνία, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συνένεση ποιοι είναι οι κοινοί ευρωπαϊκοί Γανόνε που πρέπει να υιοθετηθούν για να διευκολυνθούν οι κοινοτικέ αλλαγές, δεν φαίνεται είναι ο καλύτερο τρόπο τον οποίο έχουν αντιμετωπίσει τα πράγματα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει το νομοθετικό πλαίσιο να βελτιωθεί και προτείνουμε τα εξή. Θα πρέπει να δίδονται σαφεί πληροφορίε και ενημέρωση για το πώς η, ενημέρωση, η εναρμόνιση θα οδηγήσει σε καλύτερη ε, εφαρμογή της οδηγίας μας. Έδωσε η Επίτροπος Κούνεβα σε σχέση με το θέμα αυτό κάποιες προφορίες, αλλά πιστεύουμε ότι χρειάζεται πολλές περισσότερες. Κάποια θέματα όπως ο στόχος όσον αφορά τις ε, υπηρεσίες που καλύπτονται, πώς μπορούμε να φτάσουμε σε πλήρη εναρμόνιση, ε, τι σημαίνει αυτό για το δίκαιο της κάθε χώρας είναι απαραίτητο. Και επίσης θα πρέπει να δούμε πώς ε, τα, οι διάφορες ε, νομοθεσίες σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο, το συμβατικό δίκαιο και όλα αυτά είναι να αρμονιστούν. Κάποιο στοιχείο το οποίο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη συζήτηση είναι ότι όλοι προσπαθούμε να υπηρετήσουμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Θα πρέπει όλοι αυτά λοιπόν να εξεταστούν ως ένα ενιαίο πακέτο. Οποιαδήποτε αλλαγή γίνει στην ε, εθνική ε, νομοθεσία δεν είναι απαραίτητο κάτι το αρνητικό. Θα ήθελα κυρίως να τονίσω τρία στοιχεία τα οποία αυτή τη στιγμή κατά την άποψή μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ο μοναδικό τρόπος να έχουμε ένα πλήρως εναρμονισμένο νομοθετικό πλαίσιο και πλήρη προστασία των καταναλωτών. Γι' αυτό θα ήθελαμε να ζητήσουμε από το Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να μην αποδυναμωθεί αυτή η πλήρη εναρμόνιση την οποία τίνουμε. Όσον αφορά του τομεί στου οποίου θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση, στα πλαίσια αυτής της πρότασης. Πιστεύουμε ότι η πρόταση καλύπτει ήδη πολλές από τους, ε, πολλούς από τους ε, τομείς κλειδιά που αφορούν τις υπηρεσίες που ε, αναπτύσσουν δραστηριότητες διευθυσιακώς. αρχή της υπαναχώρησης, ενημέρωση των καταναλωτών, συνθήκες για την άσκηση αυτού του δικαιώματος υπαναχώρησης και αλλαγής άποψης του καταναλωτών νομικές εγγύσεις υπάρχουν παρόλα αυτά και άλλα θέματα τα οποία πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να εναρμονιστούν ιδιαίτερως οι συμβατικές υποχρεώσεις ε, του καθενός για την παροχή πληροφοριών. Τρίτο στοιχείο που αφορά την πρόταση, το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Συμφωνούμε ότι η πρόταση θα πρέπει να εξασφαλίσει ένα κοινό υψηλό επίπεδο προστασία των καταναλωτών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει για το ενδοησιακό εμπόριο να αισθάνονται εμπιστοσύνη οι καταναλωτέ. Θα πρέπει βεβαίω να αποφασίσουμε ποιο είναι το επίπεδο και να είναι το ίδιο επίπεδο αυτό σε όλη την Ευρώπη. Όταν συζητούμε το επίπεδο προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να επιλέξουμε το εθνικά πιο ευαίσθητο σύστημα. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα διαδικασιών που θα βασίζονται σε στοιχεία αντικειμενικά μετά από την συλλογή των κατάλληλων δεδομένων από τους ενδιαφερομένους, ώστε να υπάρχουν με απόλυτη σαφήνεια δικαιώματα και υποχρεώσεις των κατανοητών. Οι διάφορες ενώσεις καταναλωτές πιστεύω ότι μπορούν να παίξουν εδώ δια, ε, σημαντικό ρόλο για το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχουν την προστασία των καταναλωτών υψηλού επίπεδου ε, ε, στοιχεία. Τελειώνοντας θα ήθελα να ενθαρρύνω τους ε, εθνικούς ε, νομοθέτες, τους κοινοτικούς νομοθέτες και τους ε, υπεύθυνου των, κατα... των των καταναλωτών να κάνουν μία πάρα πολύ καλή συζήτηση ώστε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση win-win δηλαδή στην οποία όλοι θα είναι κερδισμένοι. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε, δεδομένου ότι πρόκειται ένα πολύ σημαντικό θέμα, να συζητήσουμε τι θετικέ συζητήσει μεταξύ μα που να καταλήξουμε σε τελικέ αποφάσει. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ που Κρατήσατε και το χρόνο που σας είχε δοθεί. Η κυρία Καρόλου Τώρα δίνω το λόγο εις ε, ε, ε στην ε, καθηγήτρια Καρόλο Μπέρντο Βενσέλ του, Πανεπιστημίου ζωμούλα. Ευχαριστώ. Ε, κυρίες και κύριοι ε, βουλευτές, ε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τους ευρωβουλευτές που μου επιτρέπουν να σχολιάσω αυτό το βασικό θέμα του ενοχικού δικαίου διότι ε, συμμετέχω σαν καθηγήτρια δικαίου και συγκεκριμένος του ενοχικού. Προφορικά βέβαια θα παρουσιάσω πολύ λίγα σχόλια και έχω υποβάλει την γραπτή μου παρουσίαση. Πρόκειται για το πρώτο εγκάρσιο κείμενο για να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς. Το κοινοτικό δίκαιο επί του θέματος είναι σε ένα βασικό θέμα και τίποτα δεν πρέπει αυτή τη στιγμή ε, να παραμεληθεί διότι πολύ σωστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επιζητεί μία συνοχή και το κείμενο αυτό θα πρέπει να είναι ανάλογο των προσδοκιών που έχει προκαλέσει. Καταρχήν θα πρέπει ε, να, να κοιτάξουμε τι είναι οι στόχοι μας. Θα μπορέσουμε να συζητήσουμε την εφαρμογή της οδηγίας η οποία δημιουργεί πολλά προβλήματα και ε, χρειάζεται μία ε, οδηγία η οποία είναι περιορισμένη. Το άρθρο 3 είναι πολύ περιορισμένο αλλά αυτός δεν είναι ο στόχος μας. Αυτό το οποίο ε, είναι ενδιαφέρον είναι ότι αυτή τη στιγμή το κείμενο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και υπάρχουν τρεις κριτικές τις οποίες μπορεί κανείς να απευθύνει. Καταρχήν πρόκειται για την ασάφεια των ενιών κλειδί οι οποίες θα περιγράψουν ε, το επίπεδο των ε, διαφόρων θεμάτων αυτών. Πρόκειται για την ε, για ε, την ε, προστασία των καταναλωτών και τέλος την πλήρη εναρμόνιση η οποία θα δώσει τη δυνατότητα να διευρύνει κανείς ή να παρουσιάσει τις πρώτες κριτικές. Το, το βασικό πρόβλημα οφείλεται στο ότι πρόκειται για μία πλήρη εναρμόνιση και ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να περιγράψουμε το πεδίο αυτό με σαφή και ακριβή τρόπο, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει τώρα. Ε, ε, ο πιο προβληματικό θέμα είναι το θέμα των πολίσεων και είναι μια βασική αρχή διότι άπαξ και καθορίσουμε τις πωλήσει θα μπορέσουμε να περιγράψουμε το πεδίο το πεδίο ισχύς της οδηγίας και ε, αυτό δεν καθορίζεται στην οδηγία. Η οδηγία περιγράφεται σαν μία, ε, στην οδηγία περιγράφεται σαν μία πώληση. Άρα άπαξ είναι πώληση, βλέπουμε ότι μία διάταξη προβλέπει ότι εφαρμόζεται το δίκαιο των πωλήσεων στα μικτά, στις μικτές συμβάσεις, δηλαδή σε συνδυασμό παροχής υπηρεσιών και πωλήσεως αγαθών. Όλα αυτά είναι πολύ ασαφή και δεν μπορούμε μπορούμε να ξέρουμε τι είναι ένα τέτοιο, κάποια τέτοια σύμβαση. Εφόσον κανείς δεν αναφέρεται σε μεταφορά ιδιοκτησίας που συνεπάγεται η πώληση, συμβαίνει ότι υπάρχει συγχρόνως κάλυψη των της παροχής υπηρεσιών. Επίσης η πώληση αναφέρεται σε αγαθά το οποίο είναι ουσιαστικά εις, το, στην οδηγία μια περιγραφή των σωματικών αγαθών πράγμα το οποίο δεν σημαίνει το ίδιο πράγμα σε όλες τις χώρες άρα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί η πώληση άρα θα πρέπει την κατάλληλη στιγμή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να μας πει τι είναι ε, ένα κινητό αγαθό για να μπορέσει να υπάρξει ένα κοινό και ενιαίο δίκαιο των αγαθών το οποίο όλοι θα επιθυμούσαμε. Μία δεύτερη κριτική την οποία μπορούμε να κάνουμε και να φέρουμε είναι η μείωση της ε, προστασίας των καταναλωτών σε ορισμένα κράτη-μέλη γιατί υπάρχει μία ελάχιστη εναρμόνιση και αυτό δεν θα δημιουργούσε προβλήματα. Αλλά επειδή υπάρχει πραγματική εναρμόνιση, γι' αυτό η μείωση ε, της προστασίας είναι ουσιαστική και θα λάβω δύο παραδείγματα, ένα ακραίο και ένα κλασικό. Καταρχήν η η ε, πώληση πρέπει να συνεπάγεται την εγγύηση συμμορφώσεως. Δεν μπορούμε δηλαδή να εφαρμόσουμε ένα πιο προστατευτικό καθεστώς και ένα εθνικό καθεστώς που να είναι πιο προστατευτικό. Εδώ θα αναφερθώ σε δύο θέματα στην εγγύηση. Η εγγύηση καλύπτει δύο χρόνια από κάποιο σημείο. Δηλαδή ε, είτε από την μεταφορά των κινδύνων είτε από την ε, ηλική ε, την ηλική παράδοση δύο χρόνια μετά την παράδοση και εάν αύριο ισχύσει αυτό το κείμενο δεν θα μπορέσουν να ισχύσουν τα πιο προστατευτικά εθνικά συστήματα και ε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα ελαττώματα μπορούν να προκύψουν μετά τα δύο χρόνια και σήμερα αυτό καλύπτεται από το πιο προστατευτικό εθνικό δίκαιο το οποίο επιτρέπει μία ελάχιστη εναρμόνιση αλλά δεν θα επιτρέψει αύριο μία πλήρης εναρμόνιση. Επίσης όσον αφορά την ε, ε, ε, μείωση της προστασίας των καταναλωτών αναφέρεται στην ιεράρχηση των ε, λύσεων. Ε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μία ελεύθερη επιλογή για τον καταναλωτή εφόσον η αντικατάσταση προέχει. Τα εθνικά δίκαια έχουν ε, πιο σοβαρές κυρώσεις, δηλαδή με την εναρμόνιση το περίεργο αποτέλεσμα θα είναι ότι ένας επαγγελματίας θα είναι πιο προστατευμένος από ότι ο καταναλωτής. Επίσης πέραν του καθεστώτος της πωλήσεως η μείωση της προστασίας του καταναλωτή οφείλεται εις ε, τις υπερβολικές ρίστες ιδίως εις την απαρίθμηση ε, των, ε, των ε, ρήτρων πλήρους εναρμονήσεως διότι η πλήρης εναρμόνιση οδηγεί στην κατάρτιση κλειστών καταλόγων και δεν θα μπορούν τα κράτη-μέλη να προσθέσουν άλλες ρήτρες υπερβολικές εις τα, τις κοινοτικές ρυθμίσεις. Υπάρχουν όμως ήδη, υπάρχει ήδη μια μαύρη λίστα που δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί διότι όλα τα κράτη-μέλη δεν ε, καλύπτονται από τις ίδιες ρήτρε. Θα πρέπει ε, στην οδηγία να υπάρχει συνένεση άρα σε πολλά κράτη θα μειωθεί η προστασία των καταναλωτών. Αλλά οι περισσότερες κρίσεις μας για το κείμενο ε, δεν θα ήταν τόσο σημαντικές εάν δεν αποβλέπαμε την πλήρη εναρμόνιση και τελειώνω με την πλήρη εναρμόνιση διότι με την νέα αυτή κατεύθυνση του ε, δικαίου των καταναλωτών είναι επικίνδυνη και ε, μία ψευδέστηση διότι ουσιαστικά αναφέρεται σε συμβατικά εγκάρσια και οριζόντια δικαιώματα και υποχρεώνει να υπάρξουν ε, στενές ερμηνείες για να οριοθετηθεί το πεδίο εφαρμογής, πράγμα το οποίο δεν είναι δυνατόν σε μία διασυνοριακή ε, συναλλαγή στην κοινότητα και επίσης θα αποσταθεροποιήσει τα εθνικά δίκαια και θα δημιουργήσει ε, συμβατότητες δικαίου εντός των εθνικών δικαίων διότι ε, θα υπάρξει μία παγωμένη παρουσίαση, δεν θα υπάρχει μία εξέλιξη και θα εμποδιστεί ε, να υπάρξει μία αύξηση της προστασίας του καταναλωτού. Επίσης υπάρχουν και ψευδεστήσεις όσον αφορά τα ευεργετήματα διότι ε, δεν θα υπάρξει μία βελτίωση της προστασίας διασυνοριακά δεν θα διότι οι καταναλωτές οι οποίοι συναλλάζονται διασυνοριακά δεν γνωρίζουν ε, τις, τα δικαιώματά τους και θα αυξηθούν οι ε, διαφορές και ε, το δικαστικό άχθος. Άρα η νομοθεσία θα πρέπει να είναι πολύ ε, συγκεκριμένη εις ε, την εφαρμογή της, παραδείγματος χάρη όσον αφορά τις προθεσμίες και να καλύπτει τους καταναλωτές περισσότερο από ότι τα πιο προστατευτικά εθνικά συστήματα. Κάτι τέτοιο επιθυμούν και οι αρχές της κοινότητος και τα κρατη και δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία που μας δίνεται να ρυθμίσουμε τον τομέα αυτό του ενοχικού δικαίου. Ωραία. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν σημαντικό αυτό το θέμα και πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις πράγματι, όχι προβλήματα. Από το Eurocommerce, κύριε Λίν, μπορείτε να μας πείτε τι θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η νομοθεσία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να σας πω της εξ πως ε, το Eurocommerce ε, και η Βρετανική Ένωση Λιανικού Εμπορίου που συνήθως εκπροσωπώ υποστηρίζει σε γενικές γραμμές αυτή την πρόταση. Και εκεί βασίζονται οι παρατηρήσεις μου. Μάλιστα εμείς θεωρούμε πως το να δημιουργηθεί μια τεράστια ενιαία αγορά ε, για τους καταναλωτές ε, που θα λειτουργεί πλήρως πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα αναμένουμε θετικά και βεβαίως μια τέτοια αγορά που θα προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών και θα υπάρχει και ανταγωνισμός παντού είναι κάτι θετικό. Μάλιστα στο τωρινό οικονομικό κλίμα θα δώσει κάποιο φως στο βάθος του τούνελ και εμείς θεωρούμε πως ε, μπορούμε να συνεισφέρουμε για την επίτευξη αυτού του στόχου γι' αυτό την υποστηρίζουμε τουλάχιστον όσο παραμένει μια ισορροπημένη και πρακτική πρόταση. Το βασικό μας μήνυμα σήμερα είναι πρώτα απ' όλα ότι εμείς είμαστε υπέρ της πλήρους εναρμόνισης ως ε, την καλύτερη μέθοδο για το πώς θα πρέπει οι καταναλωτές και οι επιχειρήσει να κινηθούν στο μέλλον. Και μάλιστα δεν θέλουμε κάποια συγκεκριμένη ε, αλλαγή και είμαστε κατά κάποιον άλλον, απλά θέλουμε να υπάρχει πλήρης εναρμόνιση γιατί θα μειωθεί το κόστος και η πολυπλοκότητα. Δεύτερον, Υποστηρίζουμε την πρόταση ως ένα ισορροπημένο πρακτικό πακέτο και όσο παραμένει πακέτο. Τρίτον, εμείς ε, δεν αναμένουμε να δούμε κάποια μείωση της σημασίας της προστασίας των καταναλωτών και θεωρούμε πως δεν κάνει κάτι τέτοιο αυτή η πρόταση ε, ουσιαστικά. Και πρέπει πάντα να θυμόμαστε πως οι επιχειρήσεις, πολλές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να προχωράνε πέρα από αυτά που ορίζει ο νόμος χωρίς να τις εξαναγκάζει κάποιος μόνο και μόνο για λόγους ανταγωνισμού και ακόμα και αν αυτή η πρόταση αλλάζει κάπως τα πράγματα αυτό δεν σημαίνει πως οι επιχειρήσεις θα σταματήσουν να κάνουν τις προσφορές ε, που κάνουν αυτή τη στιγμή όσον αφορά την προστασία των καναλτών. Τέταρτον, είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε οικοδομητικά για να εξετάσουμε και να υποστηρίξουμε συγκεκριμένες πρακτικές προτάσεις ε, αναλογικού χαρακτήρα που θα υποβληθούν για να προστατευτούν οι καταναλωτές σε όλα τα κράτη-μέλη και να αποδεχθούν αυτή την εναρμόνιση. Η έκκλησή μας είναι απλά να είμαστε ρεαλιστές όσον αφορά το κόστος για τις τιμές και τις θέσεις εργασίας τελικά. Πέμπτον, θεωρούμε πως το πεδίο εφαρμογή είναι λίγο πολύ σωστό και θέλουμε να δούμε ε, το εάν και οι υπηρεσίες ε, μπορούν να συμπεριληφθούν πλήρως και όχι μόνο εν μέρη. Γνωρίζω παραδείγματο χάρη πως κάποια άλλη κλάδη, π.χ. αυτοί προσφέρουν ταξιδιωτικά πακέτα, θα ήθελα να συμπεριληφθούν εδώ και όχι σε ένα ξεχωριστό πακέτο. Έκτον, εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες αλλαγές, να... όπως κάποιες δήματα π.χ. την πληρωμή του κόστους για κάποιες παραδόσεις ε, κατοίκων. Τώρα, Βεβαίω η ενιαία αγορά για να λειτουργήσει πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διασυνοριακών συναλλαγών και απαραίτητη εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Ο κατα... κανονισμό Ρώμη 1 δίνει αυτή την εμπιστοσύνη στου καταναλωτέ. Είναι γνωστό πω οι επιχειρήσει έχουν επιφυλάξει για αυτόν τον κανονισμό, αλλά δεν θεωρούμε πω στο πλαίσιο αυτή τη πρόταση είναι σωστό να ε- επανεξετάσουμε αυτόν τον κανονισμό. Αυτό το οποίο χρειάζονται οι επιχειρήσει όντω είναι συμβατικό δίκαιο και προστασία των καταναλωτών που θα τους επιτρέψει να κάνουν τις προσφορέ που θέλουν και να αντιμετωπίζουν τους διασυνοριακούς καταναλωτές με τον ίδιο τρόπο όπως τους εθνικούς. Έτσι θα μπορέσουν να επεκτείνουν τους ορίζοντε τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους. Πρώτον, με μια ρήτρα εσωτερική αγοράς. Δεύτερον, με την πλήρη εναρμόνιση. Από του δύο αυτού τρόπου, μόνο η πλήρη εναρμόνιση σέβεται πλήρως και τον κανονισμό Ρώμη 1 και τον ενισχύει. Οι καταναλωτές προστατεύονται από τους δικούς τους νόμους, οι επιχειρήσεις εμπορεύονται με ενιαίους κανόνες και επειδή συμβαίνει αυτό γνωρίζουν καλύτερα τις υποχρεώσεις τους και βεβαίως θα διασφαλίσουν ε, τον σεβασμό τους είτε πρόκειται για εθνικές είτε για διασυνοριακές ε, συναλλαγές και βεβαίως αυτό ακριβώ είναι που κάνει τη διαφορά για να αποφασίσουμε επιχείρηση αν θα εμπορευτεί διασυνοριακά ή όχι. Οπότε εμεί υποστηρίζουμε πλήρω την πλήρη εναρμόνιση σε αυτή την οδηγία, ειδικά εάν ισχύσει και για του καταχρηστικού όρου των συμβάσεων. Εμεί δεν θέλουμε να υπάρξουν ε, ούτε παρεκκλήσει, ούτε ένα μείγμα ελάχιστη και μέγιστη εναρμόνιση. Εμεί θεωρούμε επίση πω το πεδίο εφαρμογή είναι λίγο πολύ σωστό. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε επί αρχή μια οδηγία η οποία καλύπτει πλήρω της υπηρεσίας ε, αντί να μείνουν εκτός οι ε, εγγυήσεις. Αλλά βεβαίω πρέπει να γίνει αντιληπτό πως οι υπηρεσίε έχουν διαφορετικέ απαιτήσει από τα αγαθά. Αλλά όταν μιλάμε βεβαίως για την επαγγελματική επιμέλεια όσον αφορά την ε, παροχή υπηρεσιών και τις προσδοκίες του καταναλωτή ίσως να είναι ένας το, ένα, μια οδός που μπορεί να μας βοηθήσει να λειτουργήσουμε. Τώρα είναι πολύ πολύπλοκο το ζήτημα των ψηφιακών υπηρεσιών και είναι ατυχές το να προσπαθήσουμε πρώτα να τις προσθέσουμε και μετά να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Χρειάζονται οπωσδήποτε ξεχωριστές ε, ε ξεχωριστούς κανόνες είτε σε αυτή την οδηγία είτε σε μια μελλοντική οδηγία επίσης πρέπει το πεδίο εφαρμογή να είναι σαφέ σε σχέση με άλλα νομοθήματα. Εάν το ζητήματα όπω π.χ. το δικαίωμα επαναχώρηση όπω αυτό υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για το εάν ε, θα υλοποιηθούν τα πλεονεκτήματα της πλήρους εναρμόνισης. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι η συμπερίληψη των επανορθώσεων. Θέλουμε να υπάρχουν δηλαδή N.E.A. και συνεκτικοί κανόνες. Δεδομένου του ότι υποστηρίζουμε την πλήρη εναρμόνιση, το θέμα κλειδί είναι το επίπεδο αυτής της εναρμόνισης. Εμείς υποστηρίζουμε λοιπόν την οδηγία αυτή. Είναι ένα ισορροπημένο πακέτο. Θεωρούμε ότι είναι μια σωστή ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για επιχειρήσει και καταναλωτέ, Η προστασία των καταναλωτών βεβαίω ποτέ δεν είναι δωρεάν και ποτέ δεν είναι απόλυτη. Υπάρχει ένα κόστο και το κόστος το ευμίζονται καταναλωτέ. Υπάρχουν επιλογέ που πρέπει να γίνουν και να βρεθεί μια ισορροπία. Οπότε στόχο εδώ πέρα δεν θα πρέπει να είναι το υψηλότερο επίπεδο προστασία, αλλά ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, το οποίο θα είναι πρακτικό και θα εξορροπεί τις ανάγκες των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Θεωρούμε πως η, επιχειρη... η... η πρόταση αυτή το επιτυγχάνει αυτό. Υπάρχουν δύο στοιχεία εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο ανέφερε η κυρία Επίτροπο, η επιπρόσθετη προστασία για του καταναλωτέ, που συχνά είναι μεγαλύτερο βάρο για τι επιχειρήσει, αλλά σε γενικέ γραμμέ το δεχόμαστε αυτό, αρκεί να είναι μέρο ενό πακέτου. Το δεύτερο στοιχείο είναι η περαιτέρω προστασία για τι επιχειρήσει. Ε, όπως π.χ. το τι κάνουν οι επιχειρήσεις με αγαθά ε, επιστρεφόμενα, η δυνατότητα μείωσης της τιμής σε περίπτωση που έχουν πάθει υποστή μία τα αγαθά. Εδώ πέρα βεβαίως ε, πρόκειται για την προθεσμία των 14 ημερών. Είναι τα αναμενόμενα, αυτά τα οποία αναμένουν σε γενικές γραμμές οι καταναλωτές. Οποιαδήποτε παράταση όμως πέρα από τους έξι μήνες της διάταξης αντιστροφής του βάρους αποδείξεως θα διαταράξει την ισορροπία, αλλά μπορούμε να δεχτούμε τα δύο χρόνια ως περίοδο εγγύησης. Εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε έξι χρόνια, οπότε είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Οπωσδήποτε η Eurocommerce δεν θέλει μείωση του επίπεδου προστασίας των καταναλωτών. Αναμένουμε βεβαίως πως ε, δεν θα δεχτούν κάτι τέτοιο για καταναλωτέ και ο δικό μα στόχο εξάλλου είναι υψηλό επίπεδο προστασία των καταναλωτών σε μια ενιαία αγορά. Αλλά αν να λειτουργήσει η ενιαία αγορά, δεν μπορεί ο κάθε νόμος ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή σε κάθε κράτος μέλος να ενσωματωθεί σε μια κοινή νομοθεσία. Σημαντικό δεν είναι να μείνουν τα πάντα όπως έχουν, αλλά οι καταναλωτές να προστατεύονται από καταχρήσεις, να έχουν μια λογική μεταχείριση και να μπορούν να απευθυνθούν κάπου εάν πάντα πράγματα στραβά. Βεβαίω θα πρέπει ιδεοδό να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση και τότε τα ωφέλη για καταναλωτέ και επιχειρήσει είναι πολύ υψηλότερα. Θα πρέπει βεβαίω να γίνει μια διάκριση για του καταναλωτέ ανάμεσα στη μείωση τη πραγματική προστασία των καταναλωτών και απλά στην αλλαγή τρόπου παροχή αυτή τη προστασία. Εμεί θεωρούμε πω συμφωνούμε με τους ε, καταναλωτές. Δεν είμαστε ανταγωνιστές αλλά συνεργάτες. Γι' αυτό πολλές επιχειρήσεις έχουν εταιρικέ πολιτικές που πηγαίνουν πέρα από αυτά που ορίζει ο νόμος. Π.χ. εγγυήσεις 30 ημερών εντό των οποίων μπορεί να επιστρέψει για οποιοδήποτε λόγο τα αγαθά και να πάρει πίσω τα λεφτά. Το κάνουν αυτό για να κερδίσουν πελάτες. Οπότε όπως σας είπα, πιθανόν είναι πολλές επιχειρήσεις να συνεχίσουν εθελοντικά να προσφέρουν τις ίδιες εγγυήσεις προς έφεραν και πριν, αν αυτό επιθυμούν οι καταναλωτές τους. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε αυτά τα οποία ανησυχούν τους καταναλωτές. τους χάρη, το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για ελαττωματικά αγαθά όταν πρόκειται για προφανές ελάττωμα μετά από λίγο καιρό από την αγορά του αγαθού, αυτό το οποίο λέγεται δικαίωμα απόρριψη στο Ηνωμένο Βασίλειο και πολλά μέλη μας και η Βρετανική Ένωση ε, Λιανικού Εμπορίου θα μπορούσαν να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο για τις 14 ημέρες. Οπότε θέλουμε να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες των καταναλωτών. Τέλος να πω πως η Eurocommerce επίσης έχει κάποιες δικές ανησυχίες. Π.χ. η ανάγκη κάλυψης ε, των εξόδων μεταφοράς εάν έχει υπάρξει κάποια ε, η παναχώρηση του καταναλωτή και αν είναι ιδιαίτερα ακριβή η μεταφορά. Επίσης η ανάγκη να οριστούν κάποια αγαθά ως μη επιστρέψιμα γιατί δεν μπορούν ποτέ να ξαναπολυθούν για λόγους υγείας ή οποιονδήποτε άλλο. Επίσης κάποια εκλογήκευση κάποιων ε, εξαιρέσεων όπως ε, οι πωλήσει εξ και οι πωλήσει από πλασιά και κάποιοι όροι των συμβάσεων θα ε, Αναμένουμε βεβαίω να υπάρξουν συγκεκριμένε τροπολογίε για αυτά και άλλα ζητήματα, αλλά συμπερασματικά να πω πώ υποστηρίζουμε την οδηγία ω πακέτο και θεωρούμε πω η πλήρη αναμόνιση θα απλοποιήσει τον νόμο, θα μειώσει το κόστο και θα ενισχύσει την αγορά για καταναλωτέ και επιχειρήσει. Νομίζουμε ότι αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο και για του καταναλωτέ και για τι επιχειρήσει. Σα ευχαριστώ. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στην κυρία Γκόγιαντ από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών για να ακούσουμε και κάποιες εναλλακτικές προσεγγίσεις για την προστασία των καταναλωτών. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της ΜΠΑΚ θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διότι οργάνωσε την ακρόαση αυτή, αλλά διότι ασχολείται με την ανάλυση αυτής της πρότασης. Και πρέπει να πω ότι μας ανακουφίζει το ότι δίδεται περισσότερο χρόνο και προσδίδεται μεγαλύτερη σημασία σε αυτή την πρόταση γιατί αυτό σημαίνει μεγαλύτερη προστασία τους καταναλωτές. Επίσης, άκουσα την κυρία Κούνεβο που είπε ότι θέλει να εξετάσει η Επιτροπή ε, με άλλο μάτι <clears throat> αυτή την οδηγία. Άκουσα με μεγάλη ευχαρίστηση του συναδέλφους της ε, Commerce Europe και τους άλλους συναδέλφους να θέλουν περαιτέρω συζήτηση. Ας πάρουμε ραντεβού λοιπόν. Έχω λίγο χρόνο στη θέση μου, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θα ήθελα λίγο να τονίσω ότι θέλουμε εμείς να συζητηθεί αυτό το θέμα πιο λεπτομεριακά, όλα αυτά τα θέματα και θα είμαι πάρα πολύ γενική στις μου, είπα γιατί δεν έχω χρόνο. Η πρώτη παρατήρηση θέλω να κάνω, θα ήθελα να πιστεύω την προσοχή σας σε ένα θέμα πολύ σημαντικό σε αυτή την πρόταση. Εδώ μιλούμε για οδηγία που αναφέρει στα δικαιώματα των καταναλωτών. Περισσότερες δημόσιες δηλώσεις, οι, οι, οι διάφορες ε, μελέτες επιπτώσεων των συνοριακών ανταλλαγών είναι κάτι το οποίο αφορά τον κάθε καταναλωτή στην καθημερινή του ζωή. Ή πηγαίνει στο μικρό μαγαζάκι τη του, ή πηγαίνει στον οπτικό, ε, να αγοράσει γυαλιά για να διαβάζει ή κάνει, ε, αγοράζει μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που δεν περνούν ποτέ τα, τα σύνορα ή δεν έχουν ίντερνετ αλλά εν πάση περιπτώσει ε, αγοράζουν αγαθά και όλα τα καταναλωτικά αγαθά αφορώνται αυτό το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν κοινοί κανόνες και το βασικό θέμα είναι να ρωτήσουμε ποιες είναι οι ανάγκες όσον αφορά την ε, προστασία των καταναλωτών δεν πρέπει να συναυθούν τέτοιου είδου ε, συμβάσεις για την προστασία. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένα μέσο κοινοτικό οδηγία για να δοθούν κοινέ λύσεις στον τομέα των συμβάσεων αυτών που αφορούν την προστασία των καταναλωτών. Αλλά πιστεύουμε όμως ότι θα πρόκειται για μέσα ε, προοδευτικά, σύγχρονα, που θα βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές. Δηλαδή, βλέποντας από πού ξεκινάμε σήμερα να πάνουμε. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντική μέρη, πού μπορούμε να πάμε. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντική η ενιαία εσωτερική αγορά. Ότι υπάρχει η δυνατότητα ε, να δώσει περαιτέρω μυρίους κατανατές. Χρειαζόμαστε όμως αποδείξεις. Κοιτάξτε τη η Γενική Διεύθυνση ΣΑΚΟ που δημοσίευσε το περίφημο scoreboard πριν από μερικές εβδομάδες για να δείτε πώς λειτουργούν οι αγορές. Τι είπαν διάφοροι ε, λέγοντας ότι μετά από την πλήρη των αγορών θα υπάρξουν ωφέλη. Περιμένουμε να δούμε αυτά τα ωφέλη. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό όταν σχεδιάζεται ένα πανευρωπαϊκό μέτρο για την προστασία των κατανοητών, να δούμε ποιες είναι οι προσδοκίες των καταναλωτών πρώτα και να μην ασχοληθούμε κατά πρώτο λόγο με θέματα διασυνορικού εμπορίου. Και θα θέλαμε οι θετικέ επιπτώσει τη ολοκλήρωση αγορά να, να μην είναι κάτι που να αναφέρεται συνέχεια πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει αυτομάτως πλήρης ε, ε, ικανοποίηση των καταναλωτών όταν έχουμε πλήρη αναρμόνιση. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Εμείς τι υποδεικνύουμε από αυτού θέτος. Θα θέλαμε να κάνουμε τρεις προτάσεις. Και είναι κάτι το οποίο είπαν και οι προλαλήσαντες. Πρώτα απ' όλα παρακαλούμε θέλουμε μεγαλύτερη αποσαφήνιση των πραγματικών επιπτώσεων τις οδηγίες αυτής ε, στην καθημερινή ζωή των καταναλωτών. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει να δίδονται περισσότερες εξηγήσει. Και αυτό είναι κάτι καινούριο που ακούσαμε όσον αφορά την ε, ε, διαδραστικότητα αυτής της οδηγίας γενικότερα με τις άλλες μορφές δικαίου που διέπουν τη σχέση του καταναλωτή. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει <clears throat> να υπάρχει για τους καταναλωτές ε, η βεβαιότητα ότι καλύπτονται από το δίκαιο, από την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Διότι εάν γενικά ε, εφαρμοστεί έτσι όπως έχει το συμβατικό δίκαιο, θα έχουμε αυτό που έχουμε και σήμερα και στο μέλλον, κατακαιρματισμό της κάθε κατάστασης. Δεύτερη παρατήρηση. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να έχουμε μια πολύ καλή ανάλυση των εθνικών διατάξεων οι οποίες θα σταματήσουν να εφαρμόζονται όταν εφαρμοστεί η κοινοτική οδηγία, διότι αυτό δεν είναι καθόλου σαφές προς το παρόν. Και θα θέλαμε σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις σε κοινοτικό επίπεδο και ΙΜΚΟ νομίζω ότι ζήτησε την Επιτροπή να κάνει καλύτερη και πιο λεπτομερή ανάλυση και περιγραφή των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας που θα, θα σταματήσει να εφαρμόζεται, ώστε να ξέρει ο καθένας ποια κομμάτια της εθνικής νομοθεσίας θα παραμείνουν και ποια θα αντικατασταθούν με την κοινωτική νομοθεσία. Κάνετε τις προτάσεις σας ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία μονίμως εξελίσσεται, άρα θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη προστασία των καταναλωτών. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μείνουμε όλοι με σταυρωμένα χέρια. Υπάρχουν λύσεις τις οποίες εντόπισαν οι ερευνητές και θα πρέπει ενδεχομένως να τις λάβουμε υπόψη. Θα δώσω ένα εύκολο παράδειγμα. Στον ψηφιακό κόσμο υπάρχει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές τα προβλήματα διαλειτουργικότητας των ψηφιακών προϊόντων. Γιατί λοιπόν στον εκτενή κατάλογο των ε, πληροφοριών που πρέπει να δίδονται πρέπει την υπογραφή μιας σύμβασης να μην συμπεριλαμβάνεται αυτό. Δηλαδή, όταν πρέπει κάποιος να αγοράσει ένα ψηφιακό προϊόν, να ξέρει ποια είναι τα προβλήματα ε, διαλειτουργικότητας που μπορούν να τεθούν. Αυτό αφορά και το hardware και το software. Και ξέρω ότι και αυτή η έννοια του ψηφιακού προϊόντος επίσης είναι κάτι το δύσκολο να περιγράψουμε. Επίσης θα θέλαμε οι, αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις να κάνουν πιο φιλική αυτήν την όσον αφορά αυτά τα ψηφιακά προϊόντα. Τώρα, το επίπεδο της προστασίας σε σχέση με την ε, ελάχιστη ή, ή πολύ υψηλό επίπεδο εναρμόνιση. Είπε και η Γαλλίδα εκπρόσωπος ότι σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να κάνουμε κατάσταση να μην υπάρχει μπλοκάρισμα σε εθνικό επίπεδο. Να μην κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας εξηγήσω τη θέση μας για να το καταστήσω σαφές. Από την άποψη των καταναλωτών, το BEG, η δική μας οργάνωση πιστεύει ότι η ελάχιστη εναρμόνιση είναι η καλύτερο μέσον προστασίας των καταναλωτών. Αυτό είναι το σημείο κίνησης. Μπορούμε όμως να δεχτούμε ότι από κάποιες προϋποθέσεις πλήρης εναρμόνιση θα μπορούσε να αποτελέσει μια πιο ισορροπημένη άποψη εάν όντως έχουμε να κάνουμε με πραγματική ε, προστασία των καταναλωτών. Και μπορούμε να δεχθούμε την πλήρη εναρμόνιση πρώτα απ' όλα εάν γίνει σε πολύ υψηλό επίπεδο για να προστατεύσει τους καταναλωτές, δεν λέω στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο ως έννοια μπορεί να είναι και υποκειμενικό. Ξέρω ότι η Γαλλική το οι Γαλλοί και το Ενωμένο Βασίλειο μπορούν να συζητούν εσαΐ e ποιο είναι το καλύτερο. Πιστεύω λοιπόν ότι πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά όχι ίσω το τέλειο. Τώρα, η πρόταση ίσως δεν ήταν αρκετά φιλόδοξη. Κοιτάξτε, ποιε είναι οι εθνικές διατάξεις και ποια είναι η πραγματικότητα σε κάθε χώρα για να δείτε ποιος είναι ο καλύτερος και ο πιο δημιουργικός τρόπος να δημιουργήσετε μια σωστή βάση για την συζήτηση και όχι να είστε υπέρ της ε, παρούσης, ε, παρόντος, του παρόντος κατώτερου επίπεδου προστασίας. Δεύτερη παρατήρηση. Η εναρμόνιση, η πλήρης εναρμόνιση δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο να αφορά γενικότερα όλο το ενοχικό δίκαιο και διασυνοκά. Εκεί που μπορεί κάτι τέτοιο να είναι ε, εφικτό θα πρέπει να γίνει. Πρέπει να δούμε τον ορισμό, ποιες είναι, πώς μπορεί να υπολογιστούν κάποιες περίοδοι για λόγους ενημέρωσης και μπορούν να υπάρχουν περιφές, αλλά για κάποια θέματα δεν μπορεί η πλήρης εναρμόνιση να εφαρμοστεί. Διαφορετικά, όπως είπε και η Γαλλίδα συνάδελφος, θα πρόκειται για αυταπάτη. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό σε όλους τους τομείς. Εκεί που υπάρχουν διάφορες, ε, ε διάφορες παραδόσεις ή ιδιαιτερότητες εθνικές είναι πολύ δύσκολο να προσφέρει σε κάτι τέτοιο. Τώρα, εάν ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι προτάσεις και οι υποδείξεις που έγιναν, πράγμα το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ αισιόδοξο μέρου μας, δεν πιστεύουμε ότι θα σταματήσουν οι προκλήσεις για τους καταναλωτές. Δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε ευτυχείς. Θέλουμε οτιδήποτε γίνει στους καταναλωτές να είναι σωστό, να ενισχυθούν τα δικαιώματά μας και εδώ φτάνει η σχετική πράσινη βίβλος για αυτό το θέμα, αλλά αυτό είναι κάτι το διαφορετικό. Ευχαριστώ. Θέλω τώρα να αρχίσουμε τις ερωτήσεις. Να δώσω το λόγο στον κύριο Χέντριξ που δεν έχει ακόμη παρέμβει σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά ας δώσουμε πρώτα το λόγο σε όσους έχουν ερωτήσεις η κυρία Γκέπχαρ, ο κύριος ε, Χάρμπουρ, ο κύριος Σβάμπ και η κυρία Γόλης αργότερα κανείς άλλος αυτή τη στιγμή. Ξεκινάμε με αυτές τις τρεις ερωτήσεις. Θα παρακαλούσα τους ε, συναδέλφους να περιοριστούν σε ερωτήσεις, να μην υπάρχουν μακριά σχόλια για να έχουμε περισσότερες εναλλαγές. Η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις ομιλίες αυτές ε, με τελείως διαφορετική ποιότητα πρέπει να ομολογήσω. Η πρώτη μου ερώτηση απευθύνεται στον κύριο Αλμάρας διότι όταν τον καλέσαμε, τον παρακαλέσαμε να μας παρουσιάσουν ποια είναι, να μας παρουσιάσει ποια είναι τα, τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Δεν νομίζω ότι μας είπε ούτε μία λέξη σχετικά με αυτά και αναφέρθηκε απλώς στο κείμενο του νόμου. Θα ήθελα λοιπόν να μας απαντήσει στην ερώτηση που του είχαμε θέσει αρχικώς. Η δεύτερη ερώτησή μου, δεν ξέρω τώρα αν η κυρία Κούκμαν, η ε, Γκόγενς με συγχωρείτε, ή ποιος, αλλά αναφέρομαι στο θέμα του impact assessment, δηλαδή της ε, αξιολογήσεως των επιπτώσεων, διότι το ύψος της προστασίας των καταναλωτών τώρα διαφέρει αναλόγως ε, της νομικής ε, θέσεως των συμβάσεων που υπάρχουν. Εδώ μιλάμε για ελάχιστη εναρμόνιση, δηλαδή τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα δυνατότητα να έχουν πιο προωθημένο δίκαιο επί του θέματος Πιστεύω ότι όλοι μαζί πρέπει να έχουμε κοινά δικαιώματα γιατί αυτό θα έχει πολλά προσόντα για τους ε, πολίτες. Θα ήθελα όμως οι πολίτες στο τέλος να μην γυρίσουν να μας πούν ότι εμείς χάνουμε πολλά δικαιώματα ε, λόγω του τρόπου με τους οποίους λειτουργεί εδώ η νομοθεσία, πράγμα το οποίο ελέγχθη από πολλές πλευρές. Η κυρία Γκόγινς ας πούμε μας είπε ότι θα συμφωνούσε σε μία μία πλήρη εναρμόνιση στο ανώτατο επίπεδο και νομίζω ότι αυτό δεν είναι κακό. Ποια είναι όμως αυτή η ανώτατη εναρμόνιση, η κυρία Γκούτμαν ή η κυρία Γκόγιν, αν μπορεί μία από τις δύο να μου βοηθήσει. Νομίζω ήταν συγκεκριμένες ερωτήσεις για διάφορους. Το κύριο Χάρμπορ τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ε, ε, ομιλήσαντες και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξουν και περαιτέρω συνεδριάσεις. Η κυρία Γκόγινς μας είπε ότι ίσως θα έπρεπε να συναντηθούμε με τις επαγγελματικές οργανώσεις για να διατυπώσουμε κοινέ θέσεις οι οποίες θα ήταν σκόπιμες. Επ' αυτού θέλω να κάνω ορισμένα ερωτήματα και στον ε, κύριο Χέντριξ για τις μικρομεσαίες διότι είδαμε την πληροφόρηση από τα κέντρα καταναλωτών και η κυρία Γκούκμαν μας είπε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενδεχομένως δεν ξέρουν ποιο δίκαιο είναι εφαρμοστέο και ποια είναι τα δικαιώματα των καταναλωτών όπου ισχύουν σε περίπτωση διασυνοριακών πωλήσεων. Το, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα επηρεάσει όλους τους καταναλωτές που κάνουν οποιαδήποτε συναλλαγή είτε είναι διασυνοριακή είτε όχι και άρα περισσότερο στις εσωτερικές συναλλαγές τους όταν ε, λοιπόν καταρτήσαμε ε, την νομοθεσία για τις ε, παράνομες πρακτικές υπήρξε μία προώθηση στο δίκαιο καταναλωτών και σε εσωτερικές και σε διεθνείς συναλλαγές. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρουμε τώρα ποιο θα είναι το όφελος για τους καταναλωτές μέσα στην ίδια την αγορά τους. Το δεύτερο θέμα είναι ότι εάν πρόκειται ε, να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα το οποίο έχουμε προσπαθήσει οι διασυνοριακές ε, συναλλαγές όντως θα αυξηθούν και αυτό με οδηγεί ή στην δεύτερη ερώτησή μου που αναφέρεται ή στην εμβέλεια. Διότι ο τομέας όπου ενδέχεται να προχωρήσουν σημαντικά οι, ε, οι, οι ε, διασυνοριακές συναλλαγές ε, είναι ένα διαφορετικό θέμα σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Δηλαδή, Δηλαδή, εάν θέλουμε να εξετάσουμε τις συναλλαγές ηλεκτρονικές ή άλλες, πρέπει να δούμε εκεί όπου υπάρχουν οι περισσότερες διασυνοριακές συναλλαγές και όπως είχε πει η κυρία Γκόγεν, θα πρέπει αυτό να μας απασχολήσει περισσότερο. Αλλά διαφορετικά ε, ε, ενδέχεται αν δεν υπάρχει παρά μόνο ένα οριακό όφελος για τους καταναλωτές είναι ε, μία ερώτηση την οποία θα ίσως θα έπρεπε να εξετάσει και οι επίτροπες. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει μία βασική στρατηγική σε ολόκληρο το θέμα και μετά να προχωρήσουμε στην εμβάθυση. Ευχαριστώ κύριο Σουάμπ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαρίστως θα αναφερόμουν στην κυρία Γκογένς ε, διότι ε, είχα, είχα, ε, είπε πράγματα τα οποία ήταν διαφορετικά από αυτά που είχε πει η κυρία Γκόκμαν και τα οποία είχα ήδη ακούσει. Δηλαδή υπάρχουν ε, ε, διαφορετικές ε, εμπειρίες και δεν πρέπει να προωθήσουμε το διασυνοριακό δίκαιο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, Στη ε, Γερμανία αν υπογράψει κανείς ε, ένα έγγραφο από το ενοχικό δίκαιο η αντιμετώπιση είναι διαφορετική από ό,τι είναι στη Γαλλία. Πώς λοιπόν ε, ίσως μπορεί κανείς να προωθήσει ε, μία εναρμόνιση μεταξύ των εθνικών παραδόσεων διότι εγώ πιστεύω σε 30-40 χρόνια θα έχουμε ένα ενιαίο δίκαιο των καταναλωτών. Το θέμα είναι αν μπορούμε μέχρι τότε να διαμορφώσουμε την κατάσταση κατά τέτοιο τρόπο ώστε ε, στα πλαίσια του σχεδιασμού κανένας από τους συμμετέχοντες να μην να μην αποβλέπει μόνο ή στην ε, διευκόλυνση των επιχειρήσεων αλλά και στην καλύτερη διασφάλιση των καταναλωτών για να καλύψουμε δηλαδή ε, κάτι παραπάνω από αυτά που είχε πει η κυρία Κούνεβα και θα παρακολούσα ε, να σημειώσετε ότι πιστεύω ότι η κυρία Γκόγινς και η κυρία Γκούκμενς διατύπωσαν διαφορετικές απόψεις επί αυτού και πρέπει να δούμε πώς μπορούν να συγκεραστούν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, δεν έχω άλλες ερωτήσεις, αλλά θα κάνω μία συγκεκριμένη η οποία προέκυψε σε διάφορες παρεμβάσεις, δηλαδή ότι θα έπρεπε να υπάρχει εναρμονισμένη προσέγγιση και μετά να ε, ε, επιτρέψουμε παρεκκλήσεις και opt-out. Πρέπει λοιπόν να δούμε εάν ένα κράτος έχει καλύτερο ε, αστικό δίκαιο, εάν μπορεί να απόσχει και να καταφύγει στο εθνικό του, στην εθνική του νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή πώς θα λειτουργήσει το όλο σύστημα διότι θα δεν θα υπήρχε μία σαφής εναρμονισμένη διαδικασία εκτός και αν όλα αυτά περιοριζόντουσαν σε, συγκεκριμένους, σε συγκεκριμένα σημεία όπως παραδείγματος χάρη όπως έγινε σε άλλα προϊόντα όπως το time sharing. Ε, και όπου δεν υπάρχει καμία εθνική νομοθεσία η οποία μπορεί να αλλάξει κάτι τέτοιο και θα πρέπει να υπάρχει μία απόφαση και των 27 κρατών. Ένα άλλο πράγμα το οποίο με ανησυχεί και απευθύνεται περισσότερο στον εκπρόσωπο του Eurocommerce Εάν όντως όπως λέγονται τα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις ε, χρεώνουν διαφορετικά στις διάφορες χώρες σημαίνει ότι εάν ε, θέλω να αγοράσω στο διαδίκτυο ένα προϊόν και δω ότι είναι φθηνότερο στη Γαλλία μπορεί κάποιος να με υποχρεώσει να το αγοράσω στην Αγγλία που είναι πιο ακριβό διότι εσείς ε, κατακαιρματίζετε την αγορά κατά τρόπον ώστε να <clears throat> χρεώνουν διαφορετικές τιμές σε διαφορετικά μέρη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μακροπρόθεσμα αν ξέρω καλύτερα τα δικαιώματά μου μπορώ να έχω καλύτερες τιμές σε διάφορα μέρη. Ας ξεκινήσουμε όμως από τους πρώτους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη σειρά των απαντήσεων. Ε, ε, ο κύριος Σαλμάρες είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε που δεν αναφέρθηκα πολύ στα προβλήματα. Νόμιζα πως ε, η συζήτηση ήταν βασικά να προτείνουμε λύσεις. Προφανώς οι τομείς που θεωρούμε ότι είναι τομείς κλειδιά για την εναρμόνιση είναι πράγματι πηγές προβλημάτων και το είπαν όλοι ε, το γεγονός πως ε, η ελάχιστη εναρμόνιση που είχαμε μέχρι, ε, μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει σε πολλές νομοθεσίες και άρα σε διαφορετικές υποχρεώσεις που έχουν να εφαρμόσουν οι εταιρείε ε, ενοχλούν τι εταιρείε, το κάνουν δύσκολο το να δραστηριοποιηθούν διασυνοριακά και αυτέ αφορούν ε, τι πληροφορίε των καταναλωτών, του ορισμού. Ε, π.χ. εάν στη Γερμανία είναι κάτι αυστηρότερο από ότι στην δική σα αγορά που οφείλετε να προσαρμοστείτε. Επίση για το δικαίωμα υπαναχώρηση ή για την αστική ευθύνη. Βλέπετε είναι διαβίου ισχύει πύχη στην Ολλανδία, 60 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Οπότε υπάρχει και διαφορετική ιεράρχηση από τη μία χώρα στην άλλη. Όλα αυτά κάθισαν πιο δύσκολο και για τις εταιρείε τελικά να δραστηριοποιηθούν και το και σημαίνει και μεγαλύτερο κόστος. Δεν μπήκα σε λεπτομέρειες, αλλά μπορώ να σας αναφέρω τις ε, δυσκολίες και τις αποκλήσεις που υπάρχουν από τις εθνικές ε, νομοθεσίες. Νομίζω μάλιστα ότι τα έχει συγκεντρώσει όλα αυτά κάπου η Κομισιόν. Κύριε Γκόγενς. Πρώτα απ' όλα ξεκινήσω από την εύκολη ερώτηση για να απαντήσω τον κύριο Σβάμπ. Ο Γάλλος καταναλωτής που πάει στη Γερμανία για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο υπόκειται στο γερμανικό δίκαιο, γιατί αυτός, αυτός αναλαμβάνει το κίνδυνο. Ναι, το, το γνωρίζει αυτό ότι αναλαμβάνει κάποιο ρίσκο να πάει με δική του πρωτοβουλία. Βεβαίως, ακόμα και με την ελάχιστη εναρμόνιση θα μειωθούν αυτές οι διαφορές και δεν θα υπάρχουν πλέον τόσο ας πούμε σκάνδαλα μεταξύ κρατών μελών. Τώρα πώς να επικοινωνήσουμε με τους καταναλωτές. Το σημαντικό νομίζω είναι να δίνουμε αξιόπιστες πληροφορίες στους καταναλωτές και να μην τονίζουμε ιδιαίτερα την επίδραση που έχουν οι οδηγίες και οι κανονισμοί στους καταναλωτές. Γιατί ορισμένες φορές λέμε ότι καλύτερα είναι να πάω αναλυτή στο ίντερνετ κτλ. Αν θέλουμε πραγματικά προληπτικά να προωθήσουμε τις διασυνοριακές συναλλαγές κάνουμε το εξή. Βάζουμε την αστική ευθύνη του καταναλωτή. Δηλαδή υπάρχει διασυνοριακή συναλλαγή αλλά τοπική εγγύηση. Αλλά αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην οδηγία. Είναι κάτι που θα μπορούσε να γίνει για να βελτιωθεί. Για να απαντήσω στον κύριο Χάρμπορ και στην κυρία Γκέπχαρτ. Ε, μπορώ να απαντήσω από κοινού ποιος είναι ο ορισμός του υψηλού επίπεδου προστασίας καταναλωτών και αν προστατεύονται κάπου καλύτερα οι καταναλωτές. Δεν μπορώ βεβαίως να δώσουμε μια εύκολη απάντηση. Γιατί οπωσδήποτε η πρόταση ε, βελτιώνει κάποια πράγματα σχεδόν σε κάθε κράτος μέλος, αλλά το θέμα είναι ποια θα είναι η ισορροπία. Εγώ ως καταναλωτής από το Ηνωμένο Βασίλειο μπορώ να πω πως «Α, εντάξει, τώρα έχω 14 μέρες περίοδο υπαναχώρησης και δεν μπορεί κάποιος να έρθει στην πόρτα μου, αλλά δεν έχω το δικαίωμα απόρριψης». Πώς το ζυγίζουμε αυτό. Ή στην Ολλανδία δεν υπάρχει πλέον η διαβίου εγγύηση. Αντισταθμίζεται αυτό από τις 14 μέρες επαναχώρησης. Δεν μπορώ εγώ να πω ποιο είναι το καλύτερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Πρέπει να τα ζυγίσουν αυτά ε, οι άνθρωποι και να συγκρίνουν. Έχουν πολλά να πούν τα κράτη-μέλη μέσω του Συμβουλίου, γιατί γνωρίζουν ποια είναι η εθνική τους ε, κατάσταση και μπορούν να συγκρίνουν και να δουν τις καλύτερες ε, πρακτικές. Και οπωσδήποτε αυτό θα βοηθήσει και τον ορισμό του καλύτερου εφικτού επίπεδου προστασίας, δεν λέω τέλειου βεβαίως. Ναι, λέει η Πρόεδρος, όπως ξέρετε έχουμε, συζητήσει, έχουμε ζητήσει από την Κομισιόν να μας βοηθήσει με αυτούς τους συγκριτικούς ε, πίνακες για να δούμε τι αντίκτυπο θα έχει η νομοθεσία στα κράτη-μέλη και τι θα χαθεί στο κάθε κράτος μέλος ε, από πλευράς προστασίας. Νομίζω αυτό είναι κάτι που ετοιμάζεται. Ο κ. Χέντριξ νομίζω Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ακουστούν λίγο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις το σημαντικό αυτό ζήτημα καθώς είμαστε το 99% των επιχειρήσεων. Να σχολιάσω λίγο αυτά τα οποία είπε ο κύριος Χάρμπορ και η κυρία Γκέπχαρτ. Βεβαίως δεν θέλω να ασκήσω κριτική. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξεκινήσω από την κυρία Επίτροπο να πω πως υποστηρίζουμε την πλήρη εναρμόνιση και τον στόχο της πρότασης του τουλεχθέντος. Έχουμε δύο διαφορετικά ζητήματα νομίζω μπροστά μας. Στην πρόταση, στην όλη αυτή η συζήτηση, παραμελήσαμε τον αρνητικό αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν δείτε την αξιολόγηση αντικτύπου που έχει γίνει, ε, κυρίως ε, είχε δοθεί έμφαση, αν όχι αποκλειστικά, στις διασυνοριακές δραστηριότητες, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη πως οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και η οδηγία αυτή ισχύει και για αυτές τις επιχειρήσεις, τη συντριπτική δηλαδή πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Και βλέπουμε βεβαίω πως κατά τη σύνταξη αυτής της νομοθεσίας η πραγματικότητα και η καθημερινότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν ε, λήφθη υπόψη κατά τη σύνταξη αυτή της, οδηγία. Ε, ε, οδηγίας. Και θα αναφέρω και κάποια παραδείγματα γιατί του ζήτησε η κυρία Γκέπχαρτ. Πρώτα απ' όλα το δικαίωμα αυτό της ε, προσφυγής υπήρχε στην αρχική οδηγία κάτι τέτοιο και αφορούσε τον ε, τελικό πολιτή ο οποίος έχει αφαιθεί απέξω έξω όμως από αυτή την οδηγία και είναι κρίσιμο αυτό για τους ε, μικρούς πολιτές και εγκαταστάτες. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη πρόταση όταν ανασυνταχθεί αυτή η πρόταση ή να υπάρξει η αισθητική ευθύνη του παραγωγού. Και νομίζω σε αυτό συμφωνούν και οι λιανοπολιτές και οι παραγωγοί. Κατόπιν έχουμε κάποια προβλήματα με το πεδίο εφαρμογή και τη γενική αντιμετώπιση έτσι, της οδηγίας. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά το δικαίωμα αυτό των, της επαναχώρησης εντός 14 ημερών. Αυτό είναι πρόβλημα για τις μικρές επιχειρήσεις, ε, παραδείγματο χάρη, για τα λογιστικά τους, ε, για την αποθήκη τους, για τα τιμολόγια. Και αυτό δεν έχει σχέση με υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Αυτό οδηγεί σε ανεύθυνη συμπεριφορά των καταναλωτών γιατί θεωρούμε και νομίζω πως είναι λάθος εδώ η προσέγγιση της Κομισιόν πως ε, η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί καταναλωτή ξεκινάει έχοντας μια λανθασμένη υπόθεση ότι πάντα ο καταναλωτής είναι ο ασθενέστερος. Υπάρχουν καλοί και κακοί σε όλες τις πλευρές. Οπότε πρέπει να αναζητήσουμε μια πιο ισορροπημένη λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανέφερα λοιπόν το, μη, το τη διάρκεια της ε, περίοδου επαναχώρησης αλλά και τις ε, συμβάσεις που εκτός ε, τόπου επισκέψεων υπάρχουν επισκέψεις οποίες έχει ζητήσει ο καταναλωτής ε, κάτι το οποίο χρησιμοποιούν πάρα πολύ μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και... Ε, πραγματικά θα μας δυσκολεύσει πάρα πολύ ε, το να εισαχθεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Κυρία και ο κύριος Σουίν. Θα είμαι σύντομη Αφενός θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά τα οποία είπε η κυρία Γκογένς για το υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καναλτών. Είναι πολύ δύσκολο πράγματι να το ορίσουμε. Για να ορίσουμε το υψηλότερο επίπεδο προστασίας του καναλτή πρέπει να δούμε το πλήρες σύστημα προστασίας του καταναλωτή γιατί δεν είναι μόνο εντό αγωγικών αν θέλετε ο τομέας που εναρμονίζεται αφορά π.χ. το ενοχικό δίκαιο συνολικά της διατάξης που υπάρχουν εκεί πέρα και το πώς εφαρμόζεται κάτι τέτοιο π.χ. αν υπάρχει κάποιο δικαίωμα αυτό επαναχώρηση που υπάρχει εξοδικαστικά ή ποια είναι η διαδικασία ε, επίλυσης ε, διαφορών και βεβαίω και η διαδικασία μέσω των ε, δικαστηρίων. Τέλος να κάνω μια μικρή παρατηρήση κύριε με συγχωρείτε δεν ε, εκφράστηκα σωστά, και στην Γαλλία πράγματι οι υπογραφές είναι νομικά δεσμευτικές, αλλά η πραγματικότητα, όπως ξέρετε, διαφέρει από την θεωρία. Οι Γάλλοι είναι συνηθισμένοι έτσι, να, ε, να θεωρούν ότι δεσμεύονται όταν έχουν πληρώσει κάτι, όταν έχουν δώσει μια προκαταβολή. Οπότε συχνά αυτό δημιουργεί την εντύπωση πως δεν είναι δεσμευτική υπογραφή μου. Αλλά όπως σας είπα αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην νομική θεωρία και στην πράξη. Το ίδιο παραδείγματο χάρη έχουμε και όσον αφορά την ε, ενοικίηση. Ε, η εγγύηση βεβαίως δεν είναι για να πληρωθεί το τελευταίο νίκη αλλά συχνά δίνεται αυτή η εντύπωση και πως αυτό άρα είναι που ισχύει στο δίκαιο. Κύριε Γουίν. Ναι, κύριε Πρόεδρε, προφανώς δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω πλήρως πως ως αποτέλεσμα αυτής της οδηγίας θα υπάρχει διασυνοριακό εμπόριο αντί για να υπάρξει κάποιο, κάποια κατεύθυνση, κάποιο σε κάποιο άλλο ιστότοπο. Και υπάρχει λόγος που διαφέρουν διασυνοριακά οι τιμές, ε, είτε αφορά το κοινωνικό κόστος, ε, το κόστος απασχόλησης, ε, φορολογία κτλ. Οπότε υπάρχει λόγος για το ότι κατευθύνονται συχνά οι καταναλωτές στο site της χώρας τους. Γιατί διαφέρουν και οι νόμοι και αν υπάρξει πλήρης εναρμόνιση πράγματι θα υπάρχει ένας λόγος λιγότερος για να κατευθύνουμε μετά τους καταναλωτές στη site της δικής τους χώρας όπου ίσως είναι υψηλότερο κόστος αλλά τελικά πρέπει να, αποφασίσει, να αποφασίσει η αγορά σε ένα βαθμό γιατί αν υπάρξει μεγαλύτερος ανταγωνισμός θα υπάρξει μεγαλύτερη επιλογή από πλευρά των καταναλωτών και θα φανεί αυτό και στις τιμές και στην πρακτική καθώς κάποιος ε, διαπιστώσει πως οι καταναλωτές φεύγουν από την ιστοσελίδα του και αγοράζουν από αλλού, ίσως και αυτό θα στραφεί στο διασυνοριακό εμπόριο αντί να κατευθύνει τους καταναλωτές στην ιστοσελίδα της ε, χώρας τους. Αλλά βεβαίως απουσία νομικής ε, υποχρέωσης δεν υπάρχει κάποια εγγύηση ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, έχει προχωρήσει ο χρόνος και αν δεν έχετε κάποιες ερωτήσεις θα ήθελα να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της ακρόασης, στη δεύτερη ακρόαση. Κύριε Χάρμπορ, είχατε κάποια ερώτηση για την κυρία Επίτροπο. Κυρία Κούνεβα, θέλετε να απαντήσετε. Ναι, είχαμε μια ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Χάρμπορ και να συζητήσουμε και το θέμα αυτό. Η οδηγία αυτή αφορά όλες τις πωλήσει και ε, ηλεκτρονικών αγαθών, ε, συναλλαγές παραδείγματος χάρη στο Amazon και στο eBay. Οπότε οι υπηρεσίες δεν αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής ε, και για συμβάσεις υπηρεσιών που γίνονται ενώπιος ενωπίο σε κάποιο μαγαζί για συμβάσεις, όπως είπατε, υπάρχει υπηρεσιών κάτι το οποίο σας αφορά πάρα πολύ και για τα ψηφιακά ζητήματα. Η προστασία των καταναλωτών όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσίες ήταν κάτι που είχε αναφερθεί στο Πράσινη Βίβλο και στις διαβουλεύσεις και να σας αποκαλύψω κάτι. Εγώ έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη για το ψηφιακό περιεχόμενο και τα ψηφιακά δικαιώματα, αλλά πολύ ενδιαφερόμενη και ειδικά οργανώσεις καταναλωτών το θεωρούν πολύ σημαντικό ζήτημα, αλλά ταυτόχρονα έγινε σοβαρές ανησυχίες στις ε, επιχειρήσεις και μας είπαν πως λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος απαιτείται περαιτέρω ανάλυση. Γι' αυτό η Κομισιόν θα κάνει μία μελέτη για να βρει ποια είναι η έκταση του προβλήματος και το τι σημαίνει για τους καταναλωτές το να μην καλύπτεται το ψηφιακό περιεχόμενο. Οπότε τον Απρίλιο θα έχουμε μια διάσκεψη κορυφής των καταναλωτών, αν θέλετε, με εκπροσώπους ε, από όλες τις ε, χώρες, από όλα τα κράτη-μέλη και τα ψηφιακά ακριβώς προϊόντα θα είναι το αντικείμενό μας. Οπότε θα έχουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις, ε, τους γεωγραφικούς Είναι δηλαδή ένα θέμα που μας απασχολεί συνεχώς. Αλλά δεν νομίζω πως αυτή η συγκεκριμένη οδηγία θα μπορέσει να ενσωματώσει κάτι τέτοιο χωρίς να δυσκολέψουμε, να πάρα πολύ τα πράγματα. Αυτό νομίζω το επιβεβαιώνει και η μελέτη επιπτώσεων. Εγώ ευχαριστώ να προχωρήσω παραπέρα και να συνεισφέρω με μία πρόταση κάποιες πρακτικές ε, εφαρμογής για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Από πλευράς ε, νομικής, δηλαδή από πλευράς οδηγίας. Να ξεκινήσει τώρα το δεύτερο τμήμα της ακρόασης που αφορά συγκεκριμένα την προσέγγιση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων ε, σχετικά με την ευξημένη συνεργασία και θα κοιτάξουμε τα θέματα του Ευρωπαϊκού Ενοχικού Δικαίου, τα δικαιώματα του καταναλωτή και το κοινό πλαίσιο αναφοράς. Καταρχήν θα κάνει κάτι πρώτα σχόλια η κυρία Γόλης και μετά θα μιλήσουν οι συγητές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε εν ονόματι της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων αυτό που μας απασχολεί ε, ανέρχεται εις την εποχή όπου υπήρχαν δύο επιτροπές ε, που οι δύο επιτροπές ήταν μία όταν δηλαδή οι νομικές υποθέσεις και η εσωτερική αγορά ήταν μία και τότε θεωρούσαμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την αγορά για τις επιχειρήσεις και να αποφύγουμε τις δυσκολίες τις οποίες είχαμε με τις διαμάχες των διατάξεων μεταξύ της ε, πρώτης συνθήκης της Ρώμης και της δεύτερης. Ε, γι' αυτό και χρειάζεται ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς που να αναφέρεται σε όλο το ενοχικό δίκαιο και υπάρχει πάντοτε, υπάρχει όμως και μία πρόταση η οποία δεδομένου της οικονομικής υφέσιος ε, σημαίνει ότι ό,τι μπορεί να γίνει για να τονίσουμε την ε, ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά πρέπει να είναι σωστό και τώρα πρέπει να, ε, να δούμε τις λεπτομέρειες και να δούμε αν το σύστημα λειτουργεί στα πλαίσια του ενοχικού δικαίου είτε πρόκειται για το εθνικό είτε για το κοινό πλαίσιο αναφοράς. Όταν λοιπόν κοιτάμε και εξετάζουμε το σύνολο του ενοχικού δικαίου διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ορισμένοι έμποροι και πρέπει να αναρωτηθούμε αν και αυτοί πρέπει να ληφθούν υπόψη όσον αφορά τα δικαιώματα του καταναλωτή. Εάν δηλαδή ε, θα είναι σε μία προνομιούχα θέση ή σε μία υποδέστερη θέση διότι και αυτοί ε, είναι ένα βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επίσης, λόγω της οικονομικής κρίσης θα βλέπουμε όλο και περισσότερο ε, συμφωνίες μεταξύ των ε, καταναλωτών όπως στο eBay. Άρα αυτά λοιπόν που, που συμβιβάζονται. Γι' αυτό και πρέπει να δούμε ε, σωστά αυτή τη, τη σχέση και αν υπάρχει ένα διαφορετικό πλαίσιο του δικαίου καταναλωτών για να δούμε πού βρίσκεται και τουλάχιστον εμείς στην, Επιτροπή, ε, στην Νομική Επιτροπή προσπαθούμε να εξετάσουμε όλα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για αυτές τις πολύ χρήσιμες εισαγωγικές παρατηρήσεις. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μάρτιν Χέσελινγκ του Πανεπιστήμιου του πρώτο εμπειρογνώμονα. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όταν διάβασα πρώτη φορά την ε, πρόσκλησή σας για να κάνω σχόλια μεταξύ της πρότασης και του κοινού πλαισίου αναφοράς, η πρώτη μου αντίδραση ήταν ποια σχέση υπάρχει. Υπάρχει σχέση. Ούτε το σχόλιο της Επιτροπής, ούτε το περιεχόμενο αναφέρονταν ε, της πρώτης αυτή στο κοινό πλαίσιο Τώρα, πρέπει να πω ότι το παρόν σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο στην αρχή της ε, διαδικασίας οδήγησε βάση στην πρόταση, θέλω να πω ότι για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το κεκτημένο θα έπρεπε όντως να υπάρχει το κοινό πλαίσιο αναφοράς, ώστε να γίνει πιο συνεκτική η όλη διαδικασία. Και καταρχάς υπήρχε μεγάλη ανησυχία, διότι πολλοί πίστευαν το κοινό πλαίσιο αναφοράς θα μας ε, οδηγούσε ε, σε κάποιες ε, διατάξεις του ευρωπαϊκού αστικού δικαίου. Τώρα έχει αλλάξει η προσέγγιση της Επιτροπής. Έχει στραφεί σε κάτι ε, που αφορά περισσότερο τον Ευρωπαϊκό Κώδικα που αφορά την προστασία των καταναλωτών, μπορώ το Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που κάνουν λοιπόν την πρόταση αυτή να μοιάζει με την διαδικασία που θα μας οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός τέτοιου κώδικα ως κανονισμού. Ποιος είναι ο πρώτος στόχος και ειδικός στόχος. Να έχουμε μία διαφορετική ε, εικόνα στην ενιαία εσωτερική αγορά. Δηλαδή, Εδώ κατά πρώτο, πόλο, κατά πρώτο λόγο γίνεται ορισμός του πεδίου εφαρμογής του νοητικού δικαίου για την ε, προστασία των καρατών. Προηγουμένως αναφέρθηκαν οι ελληνικές πωλήσει και γίνεται λόγος για όλων των ειδών τις συμβάσεις τις μπορούν να συνάψουν οι καταναλωτές. Περιέχονται εδώ Λοιπόν, πρώτα απ' όλα υπάρχει το βασικό, η βασική υποχρέωση ενημέρωσης. Και είπαμε ότι θέλουμε να τίνουμε προς μεγάλη εναρμόνιση. Όπως σας είπα, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μας οδηγούν στο να πούμε ότι κάποια μέρα θα υπάρχει στην Ευρώπη ένας ευρωπαϊκός κώδικας για την καταναλωτές. Ας πούμε ότι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι αυτό της Γαλλίας. Διαφορετικό είναι το πρότυπο το γερμανικό και ξέρουμε ότι μέχρι τώρα όλα αυτά τα δικαιώματα που αφορούσαν τους καταναλωτές σε πολλές χώρες περιέχονταν στο αστικό δίκαιο και σε κάποιες χώρες θα είναι πιο δύσκολο να γίνει η προσαρμογή νέας κανόνης από τη Γαλλία. Πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι νομοθέτες θα μπορούσαν να εισαγάγουν νέα και εκτιμένα δικαιώματα σε αυτή την οδηγία για την προστασία των καταναλωτών. Και ίσως σε 10-15 χρόνια θα μπορούσαμε να έχουμε μία πιο περιεκτική, ένα πιο περιεκτικό σύνολο κανόνων που να αφορά την ευρύτερη προστασία των ε, δικαιωμάτων των κατανατών. Κάτι τέτοιο έχει όμως και επιπτώσεις. Τι σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι στην πράξη πολλές ε, αρμοδιότητες θα περάσουν από το εθνικό στο κοινοτικό επίπεδο. Γιατί θέσπιση αυτών των δικαιωμάτων. Επίσης, θα συνεισφέρει σε σαφή διαφοροποίηση μεταξύ των συμβάσεων B2B και B2C. Εάν όντως είναι έτσι τα πράγματα, το ενοχικό δίκαιο B2B θα παραμείνει σε εθνικό επίπεδο και θα αφορά και τις συμβάσεις που συνάπτονται σε εμπορικό επίπεδο, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον το εμπορικό δίκαιο θα σταματήσει να είναι μέρος του εθνικού ιδιωτικού δικαίου. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε εάν δεν θα είναι καλύτερα να ακολουθηθεί σε αυτή την ε, περίπτωση ε, το γαλλικό παράδειγμα παρά το γερμανικό όπως είπα που είναι πολύ διαφορετικό. Κατά την άποψή μου δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε υπέρ κατά κάποιου ε, δικιά σε οποιαδήποτε χώρα αλλά θα πρέπει η Επιτροπή, κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό είναι να γίνει αυτό το βήμα προς τα μπρος. Και ήδη σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να αναρωτηθείτε, θέλετε πραγματικά να έχετε έναν κώδικα συμπεριφοράς των Ευρωπαίων καταναλωτών. Αυτό είναι το σενάριο που θέλω να σας περιγράψω. Τώρα, όσον αφορά το ρόλο που μπορεί να παίξει το κοινό πλαίσιο αναφορά στην παρούσα κατάσταση των πραγμάτων, θα πω ότι στο σχέδιο δράσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα χρησιμοποιήσει το κοινό πλαίσιο αναφοράς στα πλαίσια του κεκτημένου, δεν έχει γίνει το μέχρι τώρα, αλλά ανήγγειλε επίσης η Επιτροπή ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσουν αυτό το κοινό πλαίσιο αναφοράς ως πηγή έμπνευση για την κατάθεση τροπολογιών. Ίσως τα μέρη του Συμβουλίου θα ήθελαν περισσότερο να κάνουν συγκρίσεις με το εθνικό δίκαιο το καθένα, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνει σύγκριση με το κείμενο το οποίο θα ήταν το πιο αντικειμενικά ε, ισοσκελισμένο ή ουδέτερο αν θέλετε. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είναι το κύριο μέλημά τους για την προσεχή οδηγία. Τώρα, κοιτώντας ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ πρότασης και κοινού πλαισίου αναφοράς. Στην ε, πρόταση δεν αναφέρεται το κοινό πλαίσιο αναφοράς. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο κειμένων. Πρώτα απ' όλα η δομή. Στο κοινό πλαίσιο αναφοράς το ενοχικό δίκαιο συμπεριλαμβάνεται στο ιδιωτικό εθνικό δίκαιο. Δεύτερον, στην πρόταση δεν γίνεται ο ορισμός κάποιων βασικών ενιών όπως η σύμβαση, η ζημία. Άρα πάλι και εδώ η οδηγία θα μπορούσε να βελτιωθεί εάν εμπνεότανε για περαιτέρω επεξηγήσει από το κοινό πλαίσιο αναφορά. Και βεβαίως το πιο σημαντικό είναι το επίπεδο προστασία των καταναλωτών. Το επίπεδο προστασία κανδονών στην προτινόμενη οδηγία είναι κατώτερο από ό,τι αυτό που υπάρχει στο κοινό πλαίσιο αναφορά. Έχω ένα κατάλογο παραδειγμάτων. Κάποια έχουν αναφερθεί. Η εγγύηση, η νομική εγγύηση δύο ετών, ακόμη και στην περίπτωση των πλυντηρίων ρούχων. Ένα άλλο το 38 παράδειγμα είναι ότι είναι άτυπο το δικαίωμα επαναχώρησης ενώ στην προτινόμενη οδηγία εγώ τα διάφορα, τα, το θέμα αυτό το κατάλαβα διαφορετικά, έδωσε διαφορετική άποψη η κυρία Κούνεβα, δεν αρκεί ένα email, δεν θεωρείται επαρκές η, η ιεράρχηση των διορθωτικών λύσεων επίσης είναι κάτι το οποίο αναφέρθηκε. Η κοινοποίηση ε, ενός ε, προϊόντος το οποίο είναι προβληματικό σε δύο μήνες λέγεται στη μία περίπτωση ότι σας οδηγεί σε πλήρη απώλεια όλων των δικαιωμάτων. Είπε κάτι διαφορετικό από το του θέματος η κυρία Επίτροπος. Πρόκειται λοιπόν για μία ε, νέα άποψη που θα συμπεριληφθεί στην οδηγία. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά παραδείγματα που ήθελα να αναφέρω. Κάποιο άλλο είναι το δικαίωμα ενημέρωση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνοδεύεται από αυτή την γενικότητα και από κάποια συγκεκριμένα διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα. Δεν τα βλέπουμε προς το παρόν. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά τα θέματα θα μπορούσε να αποφασίσει βάσει του κοινού πλαισίου αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αλλάξει τα πράγματα και να συνεισφέρει σε αυτό το που αναφέρθηκε προηγουμένω. Δηλαδή να κάνει αυτή την οδηγία μία οδηγία η οποία να οδηγεί σε μία κατάσταση win-win, ώστε να βγουν όλοι κερδισμένοι. Εάν αυξηθεί το επίπεδο προσθέσεων των καταναλωτών σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να είναι σε καλύτερη θέση και οι καταναλωτές και οι πολιτές να κερδίσουν, δεδομένου ότι θα να αρμονιστούν κάποια πράγματα, όντως θα έχουμε μία κατάσταση στην οποία όλοι θα είναι κερδισμένοι σε σχέση με την παρούσα κατάσταση. Τελική παρατήρηση, συνοψίζοντας. Ό,τι και να αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει συνειδητά να επιλέξει εάν όντως θέλει να έχει μία ισοσκελισμένη άποψη μεταξύ πρότασης και κοινού πλαισίου αναφοράς. ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω το δεύτερο ο ομιλητή, τον κύριο Μπούς από το Πανεπιστήμιο του Όσναμπρουκ να μιλήσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα το απόγευμα στην αρχή είπατε ότι δεν προσπαθείτε να βρείτε προβλήματα, εντοπίσετε προβλήματα αλλά να εξεύρετε λύσεις. Πρέπει όμως να αναφέρω ένα-δύο προβλήματα και θα ε, υποδείξω προς το τέλος και τις λύσεις που προτείνω. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα ήθελα να εστιάσω στην αλληλεπίδραση μεταξύ της προτινόμενης οδηγίας και του εθνικού υφισταμένου ενοχικού δικαίου και πόσο οι λύσεις ορισμένων ερευνητών μπορούν να εξασφαλίσουν μία ομαλή αλληλεπίδραση μεταξύ της οδηγίας και του εθνικού ενοχικού δικαίου. Θα σας πω λοιπόν ότι η σωστή λειτουργία της οδηγίας εξαρτάται από το πώς θα λειτουργήσει στα πλαίσια του εθνικού ενοχικού δικαίου. η ποιότητα μιας τέτοιας αλληλεπίδρασης θα είναι και το μέτρο αξιολογήσεως της προτινόμενης εναρμόνισης διότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία αποβλέπει στην πλήρη εναρμόνιση αποδεικνύει ότι είναι δυνατόν να εντοπίσουμε μικρά, ε, μικρές νησίδες ε, που χωρίς ε, τις αλληλεπιδράσεις στα πλαίσια αυτών των εισίδων αλλά κανείς δεν είναι, κανένας κανόνας δεν είναι απομονωμένος όλοι είναι μέρος ενός συνόλου όλοι βασίζονται στο εθνικό νομικό σύστημα άρα είναι αναγκαίο να εξετάσουμε το θέμα πιο ευρέως. Τι παρατηρούμε λοιπόν όταν ε, κοιτάξουμε την συνολική εικόνα στην τρίτη διαφάνεια ε, αυτό που συζητώ τώρα. Δηλαδή πώς οι κανόνες αυτοί αλληλεπιδρούν με τους, ε, μεταξύ τους διότι υπάρχουν προτάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε ε, ε, προσβάσεις προς ε, γειτονικές περιοχές και θα προεξοφλήσουν και ορισμένα αποτελέσματα που δεν θα επιτρέψουν στις χώρες να διατηρήσουν ή να εισάγουν νέους κανόνες που συνδυάζονται με το περιεχόμενο της οδηγίας. Και εδώ θα σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Το άρθρο 5 της προτάσεως έχει περιλαμβάνει έναν κατάλογο των πληροφοριών που υποχρεούνται να προσφέρονται. Ε, ένα από αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Αυτό όμως που δεν είναι σαφές είναι αν αυτό καλύπτει και τις πληροφορίες σχετικά με τις ε, ε, δυνητικές χρήσεις και τους ενδεχόμενους κινδύνους. Αν η απάντηση είναι αρνητική, και αυτό δεν καλύπτεται σημαίνει ότι ο κατάλογος του άρθρου 5 δεν επιτρέπει στα κράτη-μέρη να διατηρήσουν ε, και να επιβάλλουν τέτοια υποχρέωση πληροφόρησης. Και τι γίνεται με τη Γαλλία με την obligation de ε, renseignement ή με το γερμανικό culpa in contrahendo Δηλαδή αν υπάρχουν ασυμμετρίες τα κράτη-μέλη δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία εάν η οδηγία επιβάλλει έναν πλήρη κανόνα υποχρεώσεων πληροφόρησης. Αν η απάντηση είναι καταφατική τότε η οδηγία θα επηρέαζε πάρα πολύ το γενικό ενοχικό δίκαιο. Αν όμως είναι αρνητική απάντηση και δεν θα χρειαστεί να διατηρηθούν αυτοί οι εθνικοί κανόνες ενοχικού δικαίου, τότε η εναρμόνιση θα μπορέσει να προσφέρει επιπρόσθετες ε, ε, υποχρεώσεις πληροφόρηση σχετικά με την κούρπα in και ούτω καθεξής. Ε, αυτές είναι ορισμένες δυνητικές επιπτώσεις. Τώρα, σχετικά με το δίκαιο αγοραπολουσιών, ο καταναλωτής τώρα δικαιούται να του επιστραφεί εντός 7 ημερών το ποσόν εάν ε, δεν έχει ε, ε, δεν έχει παραλάβει το προϊόν. Και αυτό σημαίνει όχι σε 6 μέρες, σε 8 μέρες, σε 7. Τι γίνεται όμως αν θέλει να καταργήσει τη συμφωνία. Τι γίνεται στην ε, περίπτωση που υπάρχουν ποινικέ ρήτρε καθυστέρησης. Ορισμένα θέματα αναφέρονται στο άρθρο 27 αλλά το άρθρο 27 απλώς αναφέρει ε, ε, την αποζημίωση για καθυστερημένη παράδοση. Εάν λοιπόν ε, δεν έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις τότε μιλάμε για χρηματικές και μη χρηματικές αποζημιώσεις. Μιλάμε για ασφάλμα, για στενά εννοούμενη ευθύνη για αιτιολογίες, ε, για μετριασμό των ε, βλαβών. Δηλαδή τι γίνεται στην περίπτωση αυτή. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να διατυπώσει ε, δογματική, δογματικό δίκαιο για τις αποζημιώσεις το οποίο θα οδηγήσει σε μία μακρά περίοδο ε, νομικής ανασφαλείας και θα μειώσει ε, τις δυνατότητες συναλλαγών. Και τέλος, το τελευταίο σημείο θα σας ε, δώσω ορισμένες δυνητικές λύσεις. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν δυνατότητες επεμβάσεως στο ενοχικό δίκαιο, ενδέχεται να εξετάσουμε πώς μπορούν να συνυπάρχουν τα εθνικά συστήματα ενοχικού δικαίου και τα ευρωπαϊκά συστήματα ε, του δικαίου καταναλωτών. Δηλαδή να συνδυάσουμε την επιλεκτική πλήρη εναρμόνιση συγκεκριμένων τομέων όπως η δυνατότητα ε, ε, απόσυρσης, κατάργησης που μπορεί να ρυθμιστεί και ελάχιστη εναρμόνιση σε άλλους τομείς και ε, την δυνατότητα ορισμένων λύσεων που να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς. Και ε, το ηλεκτρονικό εμπόριο θα είναι ένας από τους υπόπτους ε, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτόν τον λόγω το πλαίσιο αναφοράς ε, και το οποίο θα περιλαμβάνει ένα γενικό πίνακα και θα δίνει ορισμένες δυνατότητες επιλεκτικής χρήσης εργαλείων και ένα άλλο θέμα που δεν αναφέρθηκε σε αυτή την ε, επιτροπή είναι τη δυνατότητα να έχει κανείς ένα μπλε κουβί είτε στις αγορές ε, μέσω του διαδικτύου όπου θα υπάρχουν ε, εναλλακτικές δυνατότητες αποκλεισμού ή περιορισμού είτε για την επιχείρηση είτε για τον καταναλωτή. Οπότε ε, με αυτόν τον τρόπο θα έβλεπε κανείς ε, ποιες είναι οι επιπτώσεις για τον καταναλωτή σε κάθε ηλεκτρονικό εμπόριο. Και πάλι νομίζω ότι ακούσαμε χρήσιμες παρεμβάσεις. Θα ήθελα λοιπόν ε, να ακούσουμε τώρα κάποιες ερωτήσεις. Δεν έχω κάποιον κατάλογο, βλέπω είμαστε και λίγοι. Δεν ξέρω αν η κυρία Γουόλης ε, από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θέλει να κάνει κάποιες ερωτήσει. Ο κύριος Χάρμπορ επίσης γνωρίζω. Κάποιος άλλος. Όχι. Ξεκινήσουμε με εσάς κυρία Γουόλης. Και βλέπουμε. Σας ευχαριστώ ε, πολύ για αυτές τις παρεμβάσεις που είναι χρήσιμες αλλά και δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όσα λύνουν κάποιες φορές έχω την αίσθηση πως κάνουμε κύκλους. Και εκεί στο τέλος μιλήσατε για κάποια μέσα κατ' επιλογή μήπως ε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τομεακές οδηγίες σε ορισμένους τομείς ανταυτού. Αυτό νομίζω ε, προσπαθούσαμε να αποφύγουμε, γι' αυτό ξεκινήσαμε ή σε τελική ανάλυση αν δεν γινόταν κάτι τέτοιο να περάσουμε σε κάτι που θα επέτρεπε στους καταναλωτές να επιλέξουν, στα μέρη μάλλον με συγχωρείτε, τους συμβαλόμενους να επιλέξουν κάποιο σύστημα. Οπότε εγώ ακόμα προσπαθώ να δω ποια πρόοδο θα έχουμε τελικά. Αυτό είναι περισσότερο σχόλιο βεβαίως παρά ερώτηση. Με συγχωρείτε κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που το είπατε, το είπατε εσείς γιατί και εγώ πραγματικά είχα αυτή την απορία, πως τελικά δημιουργούν περισσότερα προβλήματα παραλύσεις. Κύριε Χάρμπορ, να σας ακούσουμε και εσάς. Και εγώ παρόμοιες σκέψεις κάνω και σχέση με την συζήτηση με την κυρία Επίτροπο για το ποιες είναι οι προτεραιότητες μας και πώς θα προχωρήσουμε. Και δεδομένου του ότι θα έχουμε και λίγο περισσότερο χρόνο, πρέπει πράγματι να υπάρχει κάποια προσθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και... Με ουσιαστικό τρόπο. Μπορεί η σημερινή συζήτηση πράγματι να έχει αυτή τη ε, δυνατότητα, αλλά δεν ξέρω αν γίνεται αυτό στο πλαίσιο αυτό. Απ' την άλλη, και γνωρίζω ότι το έχουμε συζητήσει επί πολλά χρόνια και για την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, για την δυνατότητα να υπάρξει κάποια δυνατότητα προσφυγής ε, του καταναλωτή ε, και κάποιες εγγυήσει ε, στις διασυνοριακές συναλλαγές. Επανερχόμαστε σε αυτό το οποίο είχα πει νωρίτερα. Δηλαδή υπάρχει αίσθηση ότι οι καταναλωτές ενστικτοδός είναι πιο επιφυλακτικοί με τις διασυνοριακές συναλλαγές λόγω της αβεβαιότητας και άρα εάν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό πρέπει να τους βοηθήσουμε με, κάποιους, με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο χωρίς ε, να δημιουργήσουμε κάποια προβλήματα παράλληλα στην εθνική νομοθεσία. Δεν νομίζω ότι το είχε εξετάσει αυτό η αξιολόγηση της κυρίας Κούνεβα αλλά εντάξει, δεν ξέρω Νομίζω ότι απογοητεύομαι. Αν είναι να έχουμε κάποια πρόοδο πρέπει να δούμε κάποια από αυτά τα ζητήματα. Νομίζω το είχα αναφέρει και πριν πως η ιδέα του να έχουμε μια εγγύηση online στο διαδίκτυο, μια ευρωπαϊκή εγγύηση που θα είναι συνεχώς διαθέσιμη για όλες τις συναλλαγές, κάτι το οποίο θα είναι μια επιλογή που θα είχαν οι επιχειρήσεις, ίσως είναι ένας τρόπος ε, για να προχωρήσει αυτό το ζήτημα και βεβαίως θα ωφελήσει και τις ε, χώρες εκείνες όπου δεν είναι τόσο ισχυρή η προστασία να οδηγηθούν μέσω της προτίμησης που θα δείξουν οι καταναλωτές στις διασυνοριακές συναλλαγές στο να αυξηθεί η προστασία. Ναι, ίσως θα μπορούσαν να απαντήσουν οι πυρογνωμονές μας. Χαίρομαι για το ότι εσείς ε, κύριε Μπούς είπατε πως μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια επιλεκτική πλήρη εναρμόνιση σε κάποιους τομείς γιατί αυτό έχουμε κάνει πράγματι και υπάρχει κάποιος λόγος για το ότι δεν γίνεται αυτό αλλά παρόλα αυτά θέτει πάλι το ζήτημα που ακούστηκε ότι δηλαδή αν έχουμε έναν κοινό τομέα δηλαδή, αν εγώ αγοράζω κάποια συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, να ξέρω ότι έχω τα ίδια δικαιώματα στις 27 χώρες, αλλά μετά πρέπει να δούμε ποιες είναι οι άλλες πτυχές αυτής της αγοράς, αυτού του αγαθού, που μπορεί να με καλύπτει καλύτερα η εθνική νομοθεσία. Αλλά με ανησυχεί αυτό το οποίο είπε και η κυρία Γκούρκμαν, ότι σύμφωνα με τη δική τους ε, εμπειρία οι καταναλωτές δεν ξέρουν το εθνικό τους δίκαιο. Οπότε οι συζητήσεις που είχαμε στην Επιτροπή μας πράγματι μας οδηγούν στο να καταλήξουμε στο ότι πρέπει να είναι πρακτική η νομοθεσία και να ξέρουν οι άνθρωποι τελικά τι ε, έχουν, τι δικαιώματα έχουν για να μην καταλήξουμε σε κάτι το οποίο δεν θα γνωρίζουν οι καταναλωτές και θα έχει μετά τόσο πολλές ρήτρε και εξαιρέσει που δεν θα έχει κανένα πρακτικό αντίκρισμα. Οπότε όπως είπε η κυρία Βόλης, πρέπει νομίζω να ζητήσουμε λύσεις παρά να βλέπουμε ποια είναι τα προβλήματα. Οπότε να δημιουργηθεί μια κάποια βεβαιότητα, να δίνονται κάποια βασικά δικαιώματα και να υπάρξει μια βελτίωση της θέσης των καταναλωτών. Ξέρω πως και η κυρία Κούνεβα νομίζω ήθελε να, να πει κάποια πράγματα. Θα σας δώσω μετά τον λόγο. Κύριε Μπούς και Χάσιλινγκ, έχετε τον λόγο. Κοιτάξτε αυτό το οποίο είπα για την ιδέα του Ευρωπαϊκού Κώδικα καταναλωτή μπορεί να ακούσει κάποιος επικριτικό. Ε, αυτό που εννοούσα είναι το εξή. Πρέπει να έχουμε μια ιδέα για το που, που βαδίζουμε. Προτείνεται εδώ μια οδηγία που είναι τόσο διαφορετική από αυτά που είχαμε δει στο παρελθόν, ώστε είναι ένα ιδεώδες ε, πρώτο βήμα για έναν ευρωπαϊκό καταναλωτικό κώδικα και το θέμα είναι αν θέλουμε κάτι τέτοιο. Λύνει κάποια προβλήματα, ε, ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα. Ή μπορείτε να πείτε όχι δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, θέλουμε το ενοχικό δίκαιο να ρυθμίζεται το ενοχικό δίκαιο των καταναλωτών να διαχωρίζεται, να υπάγεται στο γενικότερο ενοχικό δίκαιο, να μην υπάρχει διαχωρισμό ανάμεσα συμβάσει μεταξύ επιχειρήσεων και, μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Οπότε, θέλουμε να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Διαφέρουν τόσο πολύ, δηλαδή οι μικρές επιχειρήσεις και οι μικροέμποροι διαφέρουν τόσο πολύ από καταναλωτές. Εάν κάποιο αγοράζει π.χ. υπολογιστές, έναν υπολογιστή, και το βράδυ ε, εάν είναι μάλλον με καταναλωτής ε, έχει κάποιους περιορισμούς δεχόμαστε και προστατεύεται περισσότερο από μια μικρή επιχείρηση είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Δεύτερον, συχνά οι καταναλωτές ε, δεν ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματά τους. Φυσικό είναι αυτό και φυσικό είναι πολλοί να μην ξέρουν ότι πολλά από αυτά τα οποία εμείς λέμε δίκαιο των καταναλωτών είναι γενικό ενοχικό δίκαιο. Η καταπαράδοση, η προστασία των καταναλωτών σε πολλά κρατημέλη ακόμα και σήμερα είναι γενικό ενοχικό δίκαιο. Και η οδηγία αυτή είναι ένα κρίσιμο βήμα προς, την, ε, το διαχωρισμό του από το Γενικό Ενεργικό Δικαίωμα ή όχι. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό το να μεταφερθεί αυτή η οδηγία στο δίκαιο των κρατών μελών θα οδηγήσει σε πολλά προβλήματα εάν δεν ξέρουμε το εάν ο τελικός μας στόχος είναι ένας καταναλωτικός κώδικας ή κάτι ανάλογο. αν αυτός ο στόχος δεν πρέπει να δούμε πώς θα συμμορφωθεί με το γενικό ενοχικό δίκαιο, δεν έχει νόημα. Πρέπει να ξέρουμε άρα που βαδίζουμε μακροπρόθεσμα. Και μπορεί να είναι κάτι που θα είναι θετικό ή αρνητικό σε σχέση με τον κώδικα αυτόν. Ε, δηλαδή μπορεί να πείτε δεν θέλουμε κάτι τέτοιο καθόλου. Μπορεί να θέλετε να διατηρήσετε τη δυνατότητα των κρατών μελών να ασχολούνται με να κρατήσουν αν θέλετε τις συμβάσεις ε, τις καταναλωτικές στο πλαίσιο του γενικού ενοχικού δικαίου. Δεν ξέρω αν θα επέτρεπε κάτι τέτοιο βεβαίω το 10. Θα πρέπει νομίζω να είναι διακριτά τα δικαιώματα των καταναλωτών ε, από τους καταναλωτές. Ε, π.χ. είχαμε την υπόθεση Κομισιόν εναντίον Ολλανδίας που το αποτέλεσμα ήταν ότι έκανε το δικαστήριο πως δεν θα πρέπει να μεταφερθούν τα δικαιώματα με τέτοιο τρόπο στο εθνικό δίκαιο ώστε να μην είναι εμφανές ότι είναι δικαιώματα των καταναλωτών. Οπότε από τεχνική σκοπιά είναι δύσκολο να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο η οδηγία αυτή ως γενικό ενεργικό δίκαιο παρά αυτό το οποίο είπε η κυρία Κούνεβα πως έχουν τη δυνατότητα διεύρυνσης του ε, τα κράτη-μέλη. Πρέπει να το κάνουν υπό δύο διαφορετικέ μορφές, συμβάσει μεταξύ επιχειρήσεων και συμβάσει μεταξύ ε, επιχειρήσεων και καταναλωτή. Αυτό το ζήτημα πρέπει να το δούμε τώρα. Για να έτσι, έχουμε και μία πιο μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση. Ναι, ναι, να επανέλθω σε ένα ζήτημα, λέει η Πρόεδρος. Προσπαθώ να αντιληφθώ εδώ τις, τις συνέπειες, αλλά για να έχουμε καλύτερη ρύθμιση. Εάν έχουμε τέσσερις διαφορετικές οδηγίες, οι οποίες εμένα ως καταναλωτή μου προσφέρουν διαφορετικά δικαιώματα, αναλόγως με το που αγοράζω κάτι, αν το αγοράζω στο κατόφλι ή στο ίντερνετ ή από το τηλέφωνο, έχουμε διαφορετικές επιλογές, δεν μου φαίνεται και αυτό πολύ λογικό. Θα έπρεπε να ισχύουν τα ίδια ανεξαρτήτως του πώς αγοράζω κάτι. Και είναι και ευκολότερο και για τις επιχειρήσεις να έχουν κοινέ προδιαγραφές. Οπότε λέτε ότι αντί να έχουμε μια νομοθεσία ομπρέλα αν θέλετε για τους καταναλωτές καλύτερο θα ήταν να τροποποιούσαμε κάθε ξεχωριστή οδηγία και να έχουμε μια κοινή περίοδο υπαναχώρησης. Αυτό λέτε. Όχι. Δεν λέω αυτό. Λέω, ο κύριος ε, Χουσελίνκ. Λέω ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε αυτό το οποίο αρχικά ανακοίνωσε η Κομισιόν ανάμεσα ε, γιατί αφορά ανάμεσα σε μια οριζόντια και κάθετη αναθεώρηση και μετά ξεκίνησε από μια οριζόντια αναθεώρηση και μετά το επέκτηνε επίχει στις ε, υποχρεώσεις ε, πληροφόρησης πριν την σύμβαση και μετά θεώρησε πως αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε ευρύτερους τομείς σε πράγματα τα οποία πριν ήταν σε μια κάθετη προσέγγιση Οπότε αν θέλετε πράγματι να είναι διαφορετικοί οι κανόνες πρέπει να είναι και κάθε η προσέγγιση. Ε, οπωσδήποτε είναι λογική η πλήρης εναρμόνιση αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι μια οδηγία η οποία διευρύνει το πεδίο εφαρμογή γιατί η υποχρέωση πληροφόρηση στην οδηγία δεν περιορίζεται στα τέσσερα αυτά σημεία που αφορούσαν οι παλιές οδηγίες αφορά όλες τις συμβάσεις ε, πώλησης ε, και υπηρεσιών. Οπότε εύκολο είναι μετά να προσθεθούν και άλλες υποχρεώσεις. Πράγματα τα οποία στα περισσοτερα κάτι κράτη-μέλη είναι ζητήματα γενικών ενοχικού δικαίου. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι για να συνεισφέρουμε λίγο επικοδομητικά κατά την άποψή μου τώρα τι απαιτείται στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα να βρούμε τους τομείς εκείνους όπου μπορούμε να έχουμε μια στοχευμένη πλήρη ε, εναρμόνιση. Αυτό απαιτεί μια ανάλυση, όπως αναφέρθηκε ήδη, των ε, κανόνων εκείνων που αυτή τη στιγμή επηρεάζονται από την οδηγία, από την πρόταση οδηγίας. Δηλαδή που υπάρχουν ε, αλληλεπιδράσεις μεταξύ της οδηγίας αυτής και του γενικού ενοχικού δικαίου. Π.χ. αυτό το οποίο ανέφερα υποχρεώσεις πληροφόρησης, ε, κανόνες περιαπάτησης κτλ. Οπότε πρέπει να γίνει μια λεπτομερής ανάλυση του ποια τμήματα του γενικού ενοχικού δικαίου επηρεάζονται. Εάν είναι δυνατόν να διατυπώσουμε ευρωπαϊκούς κανόνες χωρίς να επηρεάσουμε το γενικό ε, ενοχικό δικαίωμα, όπως στην περίπτωση της επαναχώρησης, καλώς. Εάν όχι, ε, έχουμε μετά το πολιτικό ας πούμε ζήτημα που πρέπει να απαντηθεί. Δηλαδή, πόσο μακριά θέλει ο Ευρωπαίος νομοθέτης να προχωρήσει και να μπλέξει με το εθνικό ενοχικό δίκαιο. Είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσει η σχέση μεταξύ της οδηγίας και του εθνικού ενοχικού δικαίου. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από τις ε, αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Υπάρχει μια υπόθεση που εκκρεμεί αυτή τη στιγμή στο ΔΕΚ. Ο ΔΕ Γενικός ε, προτείνει για το ζήτημα του. Μέχρι ποιου ε, σημείου χρειάζεται ε, η εναρμόνιση για τις παράνομες πρακτικές να επεμβαίνει στην εθνική νομοθεσία. Πιστεύω λοιπόν ότι θα δούμε πάρα πολλές περιπτώσεις παρεμφέρειας, σαν αυτή η οποία εκρεμεί αυτή τη στιγμή εάν η οδηγία εφαρμοστεί στη μορφή που έχει τώρα. Κυρία Γόλης, έχουμε ακόμη πέντε λεπτά ακόμη διερμηνία και τελειώνουμε. Θέλετε να μιλήσετε? Όχι. Ε, τότε μπορείτε να μιλήσετε εσείς αλλά έχουμε ελάχιστο χρόνο. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Δηλαδή δεν θέλαμε απλώς να ε, ε, παρουσιάσουμε προβλήματα χωρίς να προτείνουμε λύσεις, πράγμα το οποίο έγινε για τους περισσότερους παρεμβαίνοντες. Δηλαδή προσπαθήσαμε να δείξουμε ποιες είναι οι δυσκολίες που θα προκύψουν από την πλήρη εναρμόνιση που είναι μια νέα προσέγγιση. Διότι όπως πολύ σωστά είπατε πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ του να επιτρέψουμε στην εσωτερική αγορά να λειτουργήσει καλύτερα και να βρούμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο για τους καταναλωτές. Φτάνουμε λοιπόν με την μεγαλύτερη ε, επιρροή του ε, του κοινοτικού δικαίου στο ενοχικό δίκαιο στο να υπάρχουν παρεμβολές και παρεμβάσεις και στο κοινοτικό και στο εθνικό δίκαιο. Όπως ελέγχθη πρέπει να δούμε τι θέλουμε. Εάν θέλουμε να υπάρχει διασυνοριακό εμπόριο και να υποκινήσουμε τις, τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να εμπορεύονται μεταξύ τους θα πρέπει να υπάρξει ένα, ε, μία λύση. Αλλά η μόνη λύση τότε σε αυτή την περίπτωση ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να σκεφτούμε να υπάρξει μία πλήρης ε, εναρμόνιση μόνο για το διασυνοριακό εμπόριο και όχι το εθνικό εμπόριο. Οπότε στην περίπτωση αυτή για να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη οι καταναλωτές θα χρειαστεί μεγαλύτερο επίπεδο από αυτό που προσφέρει τώρα η οδηγία. Εάν όμως πιστεύουμε ότι θέλουμε να νομοθετήσουμε συγχρόνως για τις διασυνοριακές αγορές και την εθνική αγορά, προσκρούμε στα εθνικά δίκαια που είναι πιο προστατευτικά και υπάρχει ένα μπλοκάρισμα. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε καλύτερα την εναρμόνιση προς μία κατεύθυνση και όλοι θέλουμε να έχουμε καλύτερη εσωτερική αγορά αλλά και συγχρόνως προστασία του καταναλωτού και άρα το πρόβλημα είναι η γενικευμένη ε, αγορά. Οπότε ή θέλουμε να εφαρμόσουμε σε ένα τόσο ευρύ πεδίο πιστεύουμε ότι η πλήρης εναρμόνιση δεν θα είναι η σωστή λύση, θα μπλοκάρουμε και δεν θα βρίσκουμε λύσεις και πολύ φοβούμε ότι τουλάχιστον στην τωρινή μορφή δεν υπάρχουν λύσεις. Νομίζω ότι είναι ένα καλό σημείο να σταματήσουμε και θα ήθελα απλώς να σας πω ότι βρήκα πολύ χρήσιμες όλες τις παρουσιάσεις, σας ευχαριστώ διότι θέσατε τα πράγματα κατά τέτοιο τρόπο, εμείς τα είχαμε εντοπίσει μεν, αλλά εσείς μας κατευθύνατε προς την κατεύθυνση όπου θα θέλουμε να τα κοιτάξουμε πιο λεπτομερώς, είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, μπορούμε να δούμε τι αυτό σημαίνει από πλευράς εθνικού δικαίου και αν με ρωτήσετε εμένα για τη δικιά μου επιτροπή εάν θέλουμε να τρέξουμε και να δημιουργήσουμε μία ε, σύγκρουση μεταξύ εθνικού και κοινωτικού δικαίου προφανώς όχι. Θέλουμε να υπάρξει μία προστιθέμενη αξία. Διαφορετικά αν δεν το επιτυχάνουμε ε, πρέπει να αλλάξουμε τον εστιασμό του στόχου μας και να προσπαθήσουμε να δούμε ποιες θα είναι οι περαιτέρω επιπτώσεις αυτής της νομοθεσίας και να αποφασίσουμε αν θέλουμε να καν να ακολουθήσουμε αυτή την, κατεύθυνση. Θέλω να ευχαριστήσω την, ε, την Επίτροπο η οποία ε, κάθισε και άκουσε σιωπηλά όλα αυτά που λέγαμε και ελπίζουμε ότι θα σκεφτεί για να δημιουργήσει προτάσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν και πιστεύω ότι με τη βοήθειά σας θα επιτύχουμε. Ευχαριστώ όλους και για τους λίγους ποιοτικούς ε, ευρωβουλευτές που παρέμειναν μέχρι τέλους. Ε, τελειώσαμε την συνεδρία της Επιτροπής μας αυτή την εβδομάδα και σας υπενθυμίσω ότι 9 Μαρτίου θα ψηφίσουμε στο Στρασβούργο σχετικά με την οδηγία των υγειονομικών υπηρεσιών με ε, διάφορες άλλες προτάσεις και ε, θα συζητήσουμε και το σχέδιο προτάσεως του κυρίου Χάρμπουρ. Δηλαδή έχουμε αρκετά μπροστά μας. Καλό βράδυ.